Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Άσελμπρον. Υποθέτουμε ότι αυτό λέει τουλάχιστον. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο Ζωάν Άσελμπρον, ο υπουργό Εξωτερικών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, είναι εδώ εκπροσωπώντας το Συμβούλιο των Υπουργών. και θα μας ε, πει κάτι σε σχέση με τα θέματα τα οποία έχουν ε, αντιμετωπιστεί στο Συμβουλίο Υπουργών τα τελευταία χρόνια βέβαια. Ε, ήταν στο Κίεβο, στην Τυφλίδα και την Μόσχα και ίσως θα μπορούσε να επεκταθεί και στα θέματα των επισκέψεών του δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάει μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στο Κίεβο και την Τυφλίδα. Οπότε αυτά τα οποία θα μας πούν, θα μας πει ο κ. μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Έχουμε περάσει διάφορα αυτή τη βδομάδα. Υπήρξε μια συμφωνία στη Λιβύη. Υπήρξε επίσης μια συμφωνία στην Μακεδονία για μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε νέες εκλογές. Και επίσης υπήρξε πρόοδος στο θέμα του Ιράν, το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα της εβδομάδας. Βέβαια έχουμε και αρνητικά νέα από την περίπτωση της ε, Ελλάδος, ανεξάρτητα από ποια πλευρά βλέπει κανείς το θέμα. Mm. Κύριε Άσελμπορν, θα πρέπει να φύγει κατά τις 5 στις 4 ε, παρα 5 και γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε την προσπάθεια να τηρήσουμε το χρόνο αυτό που έχουμε μέχρι τις 4 και 5, όχι παρα 5, ώστε ο πρόεδρος του Συμβουλίου να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Είναι πράγματι μια μεγάλη τιμή και χαρά να σας υποδεχτούμε ως ε, πρόεδρο του Συμβουλίου, ως και Υπουργό του Λουξεμβουργού και φυσικά η κυρία Μογκερίνη δεν σε θέση να είναι μαζί μας αυτές τις μέρες, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να μας μεταφέρετε πολλά από τα θέματα που ήθελα να συζητήσει μαζί μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Έλμαρ, θα ξεκινήσω στα γερμανικά, ίσως, για να απαντήσω το ερώτημα που μου έθεσες. Η επίσκεψή μου στο Κίεβο, στην Τυφλίδα και την Μόσχα. Και να ξεκινήσω με Γνωρίζουμε ότι η διάσκεψη κορυφής της Ρήγας ήταν μια διάσκεψη κορφής όπου νιώσαμε κάποια ματέωση σε σχέση με τα θέματα της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συμφωνία αυτή σύνδεσης θα εφαρμοστεί σε τρεις χώρες τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. Ο στόχος μας θα είναι, μαζί με την Κομισιόν και έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, για τις τρεις αυτές χώρες να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και η Προεδρία μας θα οργανώσει μια συνεδρίαση προς την κατεύθυνση αυτή για να δει πώς προχωρεί η υλοποίηση αυτών των συμφωνιών. Αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο ζητήθηκε από τη γεωργιανή πλευρά και θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε συνέχεια. Για να σας ε, περιγράψουμε στην κατάσταση εν συντομία. Η επίσκεψή μου στην ε, Μόσχα, στο Τιφλίδα και, στο... και στην Ουκρανία, στο Κίεβο, δείχνουν πόσο ε, σημαντικά είναι αυτά τα οποία διαδραματίζονται τώρα στην Ουκρανία. Η δική μου άποψη είναι ότι υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία από τη Μόσχα, από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της Συμφωνίας του Μίνσκ. Και φυσικά και η Ουκρανία βλέπει τη συμφωνία αυτή όπως και εμείς. Η Μόσχα ασχολείται περισσότερο με τις παραγράφους 3, 4, 17, 18 και 23, δηλαδή τις λεπτομεριακότερες παραγράφους Ενώ για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια πραγματική κατάπαυση πυρός για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε μια πολιτική διαδικασία. Κάτι το οποίο δεν το θεωρεί τόσο σημαντικό από ό,τι φαίνεται η Μόσχα. Επίσης, μαζί με τον πρόεδρο Ποροσέγκο και την πλευρά του Κιέβου, έχουμε δύο καλές ειδήσει ίσως από την πλευρά αυτή. Πρώτον, ότι με λίγη τύχη και με κάποια προσπάθεια μπορούμε τον Ιούλιο να έχουμε μια πρώτη ανάγνωση μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης στην Ουκρανία που να περιλαμβάνει και την μεγαλύτερη αυτονομία, την αυτοδίκηση ουσιαστικά των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας. Μπορεί λοιπόν να περάσει η πρώτη ανάγνωση για το θέμα αυτό. Και υπάρχει και η ελπίδα ότι θα μπορέσει αυτός ο νόμος να έχει, αυτή η αλλαγή να έχει εφαρμοστεί μέχρι το φθινόπωρο. Αυτά είναι λοιπόν δύο ελπιδοφόρα μηνύματα τα οποία μπορώ να σας φέρω. Αυτό το οποίο επίσης είδα στο Κίεβο με τις επαφές μου είναι ότι το κυριότερο θέμα εκεί είναι ο αγώνας κατά της διαφθοράς. Η διαφθορά είναι πανταχού παρούσα σε αυτή τη χώρα το γνωρίζει πολύ καλά ο πρόεδρος Ποροσέγκο, όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν γίνονται για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και ο επικεφαλής της, Ευρωπαϊκής, της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου είπε και ο ίδιος ότι εδώ πρέπει να σπάσουν τα μονοπόλια, πρέπει να μην μπορούν να έχουν οι ολιγάρχες αυτή την οικονομική δύναμη και φυσικά θα πρέπει να έρθουν και ενώπιον τη δικαιοσύνη αυτοί που είναι εμπεπλεγμένοι σε θέματα διαφθορά για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη διαφθορά. Εγώ είμαι ότι στην ε, Ουκρανία θα πρέπει να υπάρξει και μια αποφασιστικότητα ώστε να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές πτυχές της οικονομίας ώστε να οικοδομηθεί η οικονομία επί νέων βάσεων. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, η οποία έχει αποσταθεροποιηθεί και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ε, βασική ιδέα των συμφωνιών του Μίνσκ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εν καιρό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια αλλαγή στάσης της Ρωσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Φεντερίκα Μοντε Μογκερίνη και της ε, Προεδρίας φυσικά του Λουξεμβούργου. Έχουμε ε, εγκρίνει την ε, παράταση των κυρώσεων μέχρι το 2016. Εάν δεν υπάρξει καμία ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση, κατά την άποψή μας δεν έχει νόημα να αλλάξουμε κάτι για το καθεστώς των ε, κυρώσεων. Αυτά ήθελα να φέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι στην Τυφλίδα είχα μια πάρα πολύ θετική έκπληξη γιατί είδαμε πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται μια προσπάθεια να υλοποιηθεί η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας. Είναι απαραίτητο να υπάρξει λοιπόν και η συνεργασία και η υποστήριξη με το Κίεβο και να αντιμετωπιστεί και το θέμα της Νότιας Οσετίας, όπου βλέπει κανείς πάλι τις θλιβερές ε, αυτές εικόνες που γνώριζαμε από την Ευρώπη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να υπάρχει ένα σύρματόπλεγμα το οποίο χωρίζει τους ανθρώπους μέσα σε ένα χωριό ή σε δύο γειτονικά χωριά και μπορεί μια οικογένεια να είναι χωρισμένη στα δύο. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την λεγόμενη παγωμένη σύγκρουση. Δεν θα πρέπει να τη χάσουμε από το μυαλό μας. Και έρχομαι τώρα στα γαλλικά. Όσον αφορά τη διεύρυνση, και εδώ θα επικεντρωθώ σε τρεις χώρες κυρίως. Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία. υποψήφιες χώρες με τις οποίες έχουν ανοίξει επίσημα οι διαπραγματεύσεις και οι οποίες ε, βέβαια είναι στην αρμοδιότητα της εκπεριτροπής ε, προεδρίας. Το Λουξεμβούργο είναι γνωστό για το ότι είναι ανοιχτό προς τους άλλους. Οπότε με ικανοποίηση σας εκφράζω ότι υποψήφιες χώρες θα προσκληθούν 7 φορές για άτυπες επαφές υπό την προεδρία μας. Κάναμε δηλαδή μια παραπάνω προσπάθεια από ό,τι έχει γίνει κατά το παρελθόν και αυτό θα επιτρέψει στις υποψήφιες χώρες να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο και το στυλ των συζητήσεων που γίνονται και που θα γίνουν και έγιναν μάλλον 10 και 11 Ιουλίου στο Τζάι και θα γίνουν και στη συνέχεια 23 Ιουλίου. Οι 23 και 24 έχουμε τους υπογρούς, έχουμε το Κίμης τον Νοέμβριο, την αστική πολιτική τον Νοέμβριο επίσης και η Τουρκία και το Μαυροβούνιο με τις οποίες ανοίξαμε κεφάλαια διαπραγματεύσεων, επίσης έχουν προσκληθεί στην ΕΠΣΚΟ αύριο και μεθαύριο στο Λουξεμβούργο. Η ειδική συνεδρίαση Τζάι, εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης, θα λάβει χώρα 7 και 8 Δεκεμβρίου στο Σαράγεβο. Δεύτερο τώρα εξάμενο του 2015 θα είναι πλούσιο και σε επαφή που θα έχουμε τις υποψήφιες χώρες και σε άλλα φόρα. Υπάρχει διπουργική στο ΝΟΙΕ μέσα Σεπτεμβρίου. Έχουμε υπουργική ΝΑΤΟ 2 και 3 Δεκεμβρίου, ε, ο ΕΣΕ στο Βελιγράδι, στο Παρίσι επίσης και ακόμα το Δεκέμβριο έχουμε την υπουργική στο Ναϊρόμπι. Όλες αυτές οι επαφές θα είναι ευκαιρία για να έχουμε επαφές με τις χώρες αυτές, οι οποίες θα έρχονται σε επαφή και με τη διεθνή σκηνή. Το Λουξεμβούργο τηρεί τις υποσχέσεις. Ίσως θα έπρεπε να είχα αρχίσει με αυτό, ότι στη διάσκεψη της Θεσσαλονίκης το 2003 είπαμε ότι το μέλλον των Βαλκανίων είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα σημερινά και πολιτικά πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποψήφιε χώρε πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να προχωρήσουν στο φάκελο αυτό της διεύρυνσης, γιατί οι υποψήφιες χώρες πρέπει να κάνουν πολύ σοβαρές πρόοδους προς την Ευρώπη, οδό που επέλεξαν. Αξιολογούμε λοιπόν την κάθε υποψήφια χώρα ανάλογα με τα συγκεκριμένα επιτεύγματα. Πρέπει να προωθηθούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ευημερίας και της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ήπειρό η Λουξεμβουριανή Προεδρία θα κάνει τα πάντα, ό,τι μπορεί δηλαδή, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. 28 χώρες τους θέλουν. Υπάρχει το πακέτο διεύρυνσης που θα υποβληθεί στις 14 Οκτωβρίου, το οποίο θα είναι πιο κατανοητό, πιο ευνόητο και εκεί θα υπογραμμίσουμε τα βασικά κράτος δικαίου, οικονομική διακυβέρνηση και μεταρρύθμιση της ε, κρατικής δίκησης. Αυτή είναι μια νέα μεθοδολογία που βέβαια θα εξετάσουν περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διεύρυνση θα υιοθετηθούν στις 15 Δεκεμβρίου. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος επίσης είναι πολύ σημαντικός για να διασφαλίσουμε καλές σχέσεις αποτελεσματικές με τους εταίρους μας. Η Προεδρία λοιπόν θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπου συμμετέχει η Σερβία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 7 και 8 Οκτωβρίου. Και για την Τουρκία 25 με 26 και για το Μαυροβούνιο 25 και 26 Νοεμβρίου επίσης. Τώρα ένα χώρα, Μαυροβούνιο. Εδώ νομίζω ότι η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι στην καρδιά του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη δουλειά στο κεφάλαιο 23 και στα θέματα δικαιοσύνης και ασφάλειας και ελευθερίας που πρώτη φορά συζητήθηκαν με το Μαυροβούνιο εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι τώρα το Μαυροβούνιο προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα φαίνεται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα θέματα. Εδώ τη δυναμική αυτή πρέπει να την εγγράψουμε και στα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης. Το Λουξεμβούργο χαίρεται που έχουν ανοίξει τέσσερα νέα κεφάλαια υπό τη Λετωνική Προεδρία. Οπότε τα κεφάλαια τα οποία έχουν ανοίξει είναι 20 σήμερα. Ελπίζω τα επιπλέον κεφάλαια, μάλλον ελπίζω ότι και επιπλέον κεφάλαια θα ανοίξουν μέχρι τα τέλη του 2015. Εμείς θα διευκολύνουμε κάθε συζήτηση στο Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση βάσει βέβαια της αρχής της ομοφωνίας. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί στο ίδιο το Μαυροβούνιο, ιδιαίτερα στο τομείς κλειδί όπως είναι το κράτος δικαίου. Θέλω να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχει ευθυγραμμιστεί 100% το Μαυροβούνιο όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Είναι πραγματικά υποδειγματικό. Σερβία. Η Προεδρία είναι πεπισμένη ότι είναι θετικό να ανοίξουν για τη Σερβία τα δύο κεφάλαια για το κράτος δικαίου και για τα θέματα της ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης, 23 και 24 δηλαδή, να ανοίξουν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα κεφάλαια όταν θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το διάλογο Βελγραδίου-Πρίστινα και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει επαρκής πρόοδος για να ανοίξει και το κεφάλαιο 35. Η Προεδρία ελπίζει ότι θα μπορέσουν να, λήξουν, να ανοίξουν σύντομα και άλλα κεφάλαια υπό τη δικιά μας Προεδρία, υπό την επόμενη. Είμαστε πάντως έτοιμοι να διευκολύνουμε κάθε συζήτηση στο Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση, τηρώντας πάντα την αρχή της ομοφωνίας. Ιδίω για το κεφάλαιο 32, που είναι για τον οικονομικό έλεγχο. Εδώ ελπίζουμε ότι γρήγορα θα μπορέσει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Πάντως, η επιτυχίες της Προεδρίας μας δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των κεφαλαίων που θα μπορέσουμε να ανοίξουμε. Δεν μετριέται έτσι η επιτυχία μιας Προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει υπόψη της ότι το 2015 θα έχει πετύχει αν η Σερβία προσεγγίσει ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προδιαγραφές της, τα κριτήριά της. Αν οι Σέρβοι πολίτες έχουν μια πραγματική προοπτική να υποφεληθούν από αυτή την προσέγγιση, αν λοιπόν γίνει πιο κανονική η κατάσταση στις σχέσεις Σερβίας και Κωσυφοπεδίου και αν η περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια ενισχυθεί προς όφελος βέβαια της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των διαφερόμενων λαών. Το Συμβούλιο Σταθερότητας και Σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση Σερβία προβλέπεται για τα τέλη της χρονιάς αυτής. Θα επιτρέψει να κάνουμε έναν απολογισμό των σχέσεών μας. Η ημερομηνία δεν είναι ακόμα γνωστή. Τώρα μετά τις εκλογές της 7ης ε, Ιουνίου στην Τουρκία περιμένουμε πληροφορίες για μια νέα τουρκική κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να αναλάβει μέσα στις επόμενες 45 μέρες προκειμένου επικοδομητικά και με ρεαλισμό να συζητήσουμε την ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Τώρα προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα τους εταίρους μας σε μια περιοχή με πολύπλοκα δεδομένα, η Προεδρία αποφάσισε να οργανώσει την εξάμεινη αποστολή της ομάδας εργασίας της στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο. Συνεχίζεται επίσης η διαδικασία ένταξης. Είμαστε πεπισμένοι ότι είναι ζωτική σημασία προκειμένου η Τουρκία να βρεθεί πιο κοντά στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια δυναμική που έχουμε κερδίσει τον τελευταίο καιρό, αν μπορώ να το πω έτσι, στην διαδικασία για παράδειγμα, υπάρχουν οι υποπιτροπές οι οποίες τρία χρόνια δεν δούλευαν και τώρα συνεχίζουν τις εργασίες τους. Μετά την διαπραγματευτική στάση της Τουρκίας για το κεφάλαιο 17 για την οικονομική και νομισματική κατάσταση. Η Προεδρία θέλει μέσα στους επόμενους μήνες να προχωρήσει στο κεφάλαιο αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν στην Τουρκία όσον αφορά το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι δικές μας εργασίες πρέπει να λάβουν υπόψη μας τις πρόοδους αυτούς τους τομείς. Η Λουξεβουριανή Προεδρία επίσης εκφράζει την ικανοποίησή της που συνεχίζονται οι συνομιλίες και στην Κύπρο από τις 15 Μαΐου που ξανάρχισαν. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ θετική δυναμική μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες, να κάνουν προσπάθειες για να βρεθεί επιτέλου μια λύση διαρκείας. Ελπίζουμε όλα αυτά να δώσουν νέα πνοή στις συνομιλίες για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εξυπηρετήσει και τις δύο πλευρές. Η Προεδρία παρακολουθεί επίσης τις εργασίες της Κομισιόν όσον αφορά το διάλογο για να καταργηθεί υποχρέωση θεωρήσεων, βίζα και για να προχωρήσουν στην Τελωνιακή Ένωση. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν επί της Προεδρίας μας. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για να προωθήσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, με τη Σερβία και με το Μαυρομούνιο αυτό το εξάμεινο. Τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα πιο σημαντικά εφόσον όντως συνεργαστούμε καλά. Εδώ και μήνες το Λουξεμβούργιο είναι σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να οργανώσουμε καλά τη συνεργασία μεταξύ μας για το εξάμεινο αυτό. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται άμεσο συντονισμό ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ώστε το ευρωπαϊκό μήνυμα να περάσει με μία φωνή και αποκτά και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στη διεθνή σκηνή. Γιατί προς τα έξω. Δεν υπάρχει η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, οι μέλη, όχι. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν που μαζί και με τους συνεργάτες μου έχουμε τέτοια στενή συνεργασία, ρεαλιστική και καρποφόρα, ελπίζω, και στο μέλλον. Και με αυτό θα ολοκληρώσω, αλλά κάτι ακόμα, Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ δύο παλιούς συναδέρφους, τον κύριο Κούκαν, Έντουαρτ, και τον κύριο Βάγγελ, και τον κύριο Χόιλ. Οι οποίοι... Α, να, Έντουαρτ. 14 προς 15 Ιουλίου κατάφεραν να βγάλουν από το αδιέξοδο την κρίση, θα έλεγα, στην ε, τέως Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η δουλειά που κάνατε, το έργο σας, η κυβέρνηση θα παραιτηθεί στα τέλη της χρονιάς, ο Πρωθυπουργό επίσης, θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση για να προετοιμάσει τις εκλογές οι οποίες θα λάβουν χώρα πότε 24 Απριλίου του χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία. Αυτά πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο ο κ. Χάουιτ έχει δύσκολο Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας στο Σεράγεβο, λέει ο πρόεδρος. Στα Σκόπια εννοεί. Και ο κύριος Κούκαν επίσης. Αλλά ο κύριος Βάγγελ δεν είναι εδώ. Γιατί τι να σας πω, πού να αντέξει αφού όλη τη νύχτα έγιναν αυτές οι συνομιλίες. Ακριβώς όπως είπατε, έτσι είναι η κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πάρα πολύ ε, δύσκολη ήταν εκεί η αποστολή μας. είχε καταρρεύσει η εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, μερών και χρειάστηκε δυναμική διπλωματία για να μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα. Οπότε και έτσι προσκληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε αυτές τις προσπάθειες. Κοινοβουλευτική διπλωματία. και χωρίς να περιευθολογούμε νομίζω ότι συμβάλαμε. Ήταν πέντε ολόκληρη 24 ώρες που προσπαθούσαμε να διαμεσολαβήσουμε τελικά πάσαμε τη συμφωνία. Οπότε βέβαια χρειάζεται η προσοχή της διεθνούς κοινότητας, χρειάζεται η διεθνική πίεση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει το θέμα. Νομίζω ότι συγκρατήσαμε την κατάσταση από το να περιπέσει την καταστροφή. Οπότε είμαστε σε συνεχή επαφή με του δημοτικού εκπροσώπους μας στα Σκόπια και το Συμβούλιο οπότε θα παρακολουθεί γιατί είναι πολύ σημαντικό. και για όποιους δεν έχουν παρακολουθήσει τα τεκτονόμενα έγινε και τρομοκρατική επίθεση. Θα μπορούσε να είναι εθνοτικά τα ελαττήρια. Είχαμε 30 νεκρούς στο μου. Δεν ξέρω ίσως αυτό δεν είναι ακριβές. Ήταν τρομερό το σκηνικό. Εκεί σβήναν τη φωτιά όλο το βράδυ, ξέρετε. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να δούμε πώς κυρία Σελμπον θα υπάρχει κάποιο μέλλον για αυτή τη χώρα. Και ο κύριος Χάν μίλησε εκεί και είπε ότι θα πρέπει και η Ελλάδα να βοηθήσει ώστε να ε, κινηθεί η χώρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίω και δεν φταίμε εμεί για όλα αυτά τα φοβερά που είναι εκεί, αλλά είμαστε υπεύθυνοι για το πώ θα λάβει σωστή κατεύθυνση η χώρα. Βέβαια αυτά τα λέει μία προεδρία μετά την άλλη, τα λέμε τόσα χρόνια. Αλλά θα πρέπει κανεί με καλή πίστη να προσπαθήσει. Και ελπίζουμε να είναι σωστή η εισήγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο και να αναλυθεί η δράση στο Συμβούλιο. Τώρα, έχω ερώτημα για την Τουρκία υπάρχει και τώρα μια ευκαιρία μετά τις εκλογές δεν λέω τίποτα για τα αποτελέσματα αλλά νομίζω τώρα ξανοίγεται μια ευκαιρία Α πούμε τα πράγματα τώρα είναι πιο ρευστά υπάρχει τώρα μια μεγαλύτερη ευκαιρία για την ευρωπαϊκή διπλωματία ελπίζουμε ότι θα εκμετρηθείτε, τέλο πάντων αυτή την ευκαιρία και μια σύνδεση του Κοινοβουλίου. Εκεί τώρα καθρεφτούνται στη σύνδεση του τα προβλήματα τα αστυνομικά και άλλα. Και τέλος, κάτι άλλο το οποίο μας ανησυχεί στα Βαλκάνια, είναι η αποσταθεροποίηση, το τι γίνεται προς Ανατολάς και δεν θα πρέπει να βρεθούμε προέκπληξη. Τι θα γίνει σε ορίζοντα ενός ή δύο τριών ετών με τις χώρες που δεν τους έχουμε δώσει κάποια προοπτική σύνδεση Θα πρέπει αυτό να το πείτε στο Συμβούλιο. Οπότε να μην λέμε πώς έγινε και χάσαμε αυτές τις χώρες, να μην το λέμε αυτό σε μια τριετία. Αν τώρα κάτι κάνουμε μπορεί αυτός ο κίνδυνος να αποτραπεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κούκαν. Καλώς ήρθατε, κύριε Άσελμπρομ. Για μένα ο Ζαν Ασελμπρόμ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα συνέχειας, σταθερότητας και αξιοπιστίας. Δεν το λέω μονάχα ως κοπλιμέντο, τον ξέρω πολύ καλά και με κάποια υπερβολή ίσως θα έλεγα ότι είναι πολύ τυχερή η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σε αυτή τη χρονική στιγμή την Προεδρία του, του Συμβουλίου του Λουξεμβούργου. Εμπειρία και επαγγελματική ικανότητα, αυτό θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν πρέπει να το δείτε σαν κομπλιμέντο, είναι μια πρόσθετη ευθύνη. Όλοι περιμένουν από εσά να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση και ελπίζω και η δική σας προεδρία θα είναι πράγματι χρήσιμη για να πετύχουμε την πρόοδο που όλοι χρειαζόμαστε για να βγούμε από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Για τη Μακεδονία μοναχα μία λέξη. Δύσκολο να γίνει αυτή η συμφωνία, ήταν ένα μικρό θαύμα θα είναι εξίσου μεγάλο, μεγάλο, μεγάλη δυσκολία η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Πρέπει όλοι λοιπόν να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και να βάλουμε ένα μεγάλο μεγεθυντικό φακό στις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθούν. Λυπάμαι που άργησα, δεν άκουσα όλα τα εισαγωγικά σας λόγια, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπατε για την περιοχή των Βαλκανίων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που θα δώσετε την πρέπουσα σημασία στην μελλοντική διεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Βαλκανίων, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία δηλαδή, μπορεί κανείς να βρει και λόγους ε, απεσιοδοξία στην περιοχή άμα το θέλει. Αλλά αν είναι κανείς αισιόδοξο μπορεί να βρει πολλά επιχειρήματα υπέρ της αισιοδοξία. Η περιοχή όμως αυτή απαιτεί σαφείς αποφάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι βασιζόμαστε στη διαδικασία της ε, πρόοδου προς την ε, ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα κάνουμε εκτόσει, αλλά όταν πετύχουν αυτά που, τα, που ζητάμε από αυτού, θα πρέπει να τύχουν αναγνώριση και από τη δική μα πλευρά. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα πετύχετε στο ρόλο σα και σα εύχομαι φυσικά και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, Καλώ ήλθατε και στην Επιτροπή μα. Συγχαρητήρια για την ε, προανάληψη της Προεδρίας από το Μεγάλο Δουκάτο. Θέλω να κάνω μερικές σκέψεις για τη διεύρυνση. Όπως είπατε προηγουμένως, είχαμε κάπως ε, αρνητικές εντυπώσεις στην αρχή της θητείας αυτής μετά από τη δήλωση ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος για τη διεύρυνση τα επόμενα πέντε, τώρα τέσσερα χρόνια. Η στάση σας τώρα για το θέμα αυτό φαίνεται να έχει κάπως αναζωογονηθεί και να έχει γίνει πιο θετική ή όχι. Δεύτερον, θα μπορούσατε να μας πείτε και κάτι για τις απόψεις σας, για αυτό που αισθάνεστε σε σχέση με τις πρόσφατες διπλωματικές ενέργειες της Σερβίας που οδήγησαν στην αποτυχία του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Σρεβέντσα. δεν είναι, είναι ένα θέμα αστοχίας και της δικαιοσύνης από κάποια άποψη αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ο Ζων Άσελμπρον εξακολουθεί να είναι ο πρίτανης των Υπουργών Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η δεύτερη φορά που προεδρεύεται του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Έχω δύο ερωτήματα, δύο σχόλια ενδεχομένω. Το πρώτο ερώτημα αφορά την τρομερή καταστροφή του προηγούμενου ε, καλοκαιριού. Θυμάστε την κατάρριψη του mah 217 του αεροπλάνου της Malaysian Airlines, το οποίο κατερρίφθη. Οι πρώτες έρευνες ίσως μπορούν να μας πούν ποιος είναι υπεύθυνος για την κατάληψη αυτή και ίσως το αποτέλεσμα, τα πορίσματα αυτής της έρευνας μπορεί να δημοσιευτούν τώρα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Αν δείξουν οι έρευνες ποιος ήταν ο ένοχος για την τραγωδία αυτή, τι είδους ενέργειες μπορεί κατά την άποψή σας η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρώντας σε, αυτήν την, ε, σε αυτά τα πορίσματα. Το δεύτερο ερώτημά σα. Αναφέρατε στο πρόγραμμα της Προεδρίας του Λουξεμβούργου ότι είναι στόχο σας να ενισχύσετε την Προεδρία, της, την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο στερέωμα και βλέπω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό το δίκτυο των πρεσβειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το στόχο αυτό. Τι βλέπετε να γίνει εκεί και υπάρχει υπάρχει το εκρεμές θέμα της προξενικής αρρωγής από τις αντιπροσωπείες των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παροχής βοήθειας σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Θα μπορούσε λοιπόν αυτές οι προξενικές αντιπροσωπείες να είναι τμήμα του δικτύου των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άσεμπρομ και από μένα κάθε ευχή για την επιτυχία σας στο εξάμεινο που θα ακολουθήσει και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το πρόγραμμα εργασίας του Λουξεμβούργου που μας παρουσιάσατε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στην αρχή της ομιλίας σας, όταν μιλήσατε για την Ουκρανία. Και εσείς ήσασταν πρόσφατα στην Ουκρανία φυσικά και έχετε δει τα προβλήματα που, που συνδέονται με την διαφθορά, με την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, με την αναθεώρηση του συντάγματος. Έχουμε ακούσει πάντα ότι αυτό θα γίνει, θα προχωρήσουμε και τα λοιπά, αλλά είναι πολλά χρόνια που τα ακούμε αυτά. Θα ήθελα όμως να θέσω και ένα άλλο ερώτημα για το θέμα της ε, μείωσης του κουρέματος του χρέου της ε, Ουκρανίας. Ξέρετε σε ποιο βαθμό θα προχωρήσει αυτό, σε τι στάδιο βρίσκονται αυτέ οι διαπραγματεύσει γιατί αυτό συνδέεται και με τα προβλήματα που αναφέρατε, μεταξύ των οποίων και το θέμα της διαφθοράς. Και επίσης, εν ώψη της συζητήσεως που κάνουμε με την Ελλάδα, όπου ένα κράτος μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτήν την προσφορά, να γίνεται και σε αυτό αυτή η προσφορά που έχει γίνει για την Ουκρανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ. Συμπαθάτε με που άργησα, λέχα τον πρώτο μου τριμερή διάλογο ε, και αυτός δεν χάνεται με τίποτα. Τα συζητήσαμε χθε και θα τα ξέρετε, δεν, θα σας κλείξω. Για πέστε μου, τι σχεδιάζει η Λουξεμβουργιανή Προεδρία για το Κόσοβο και για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, γιατί έχουμε το θέμα της ε, Συμφωνίας Σταθεροποίησης. Είναι δυνατόν αυτή η υπόθεση να προωθηθεί και να το ολοκληρώσει το πρόβλημα μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Υπάρχουν προβλήματα εκεί. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο τέλος από ό,τι φαίνεται. Λένε οι ειδήσει ότι υπάρχει μια πρόοδος της διαμαντεύσης για το Κυπριακό. Μπορεί κάτι να πετύχει η διπλωματία, μπορεί να παίξει κάποιο θετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Ο επόμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε να τα πούμε. Έχω κάποιες ερωτησούλες. Θίξατε το ζήτημα της Ουκρανίας και θα ήθελα να μου πείτε τι λέτε για τον ορισμό του κ. Σακασβίλη ως κυβερνήτου της διοικητικής περιφέρειας της Οδυσσού. Μήπως αυτό θα προκαλούσε ακόμα περισσότερες ε, προστριβές στην περιοχή ή θα είναι θετικό. Επίσης, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την διεύρυνση Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για το τι γίνεται ε, με την Βοσνία. Είδατε είχαμε αυτές τις ταραχές, αυτά τα επεισόδια ε, στην εκδήλωση για την Σρεμπρένιτσα. Τι λέτε, μήπως αυτό θα έχει ε, επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Αλλά φυσικά και για τις σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας υπάρχει κίνδυνος για δυσμενή συνέπειες. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προβλέπετε για αυτό το εξάμεινο για την εντολή σας. Γιατί ο κ. Γιούνκερ στην αρχή της εντολής της Επιτροπής είχε πει ότι θα συνεχίσουμε, θα προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα γίνει κατά την εντολή μου διεύρυνση. Συμφωνείτε με την τοποθέτηση αυτή του κ. Γιούνκερ. Α, γιατί κάτι είπατε για το Μαυροβούνιο. Μήπως θα μπορούσε να επιτευχθεί η διαδικασία και έτσι να γίνει πριν το τέλος της εντολής ε, άλλη διεύρυνση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Πρέπει να χαίρεστε που διάλεξε την ε, Οδυσσό και όχι την περιοχή της Βενετίας ο κύριος Ακιασβίλη λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Άγιος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευτυχώ δεν αναφέρατε το Βίλνιου σαν υποψήφια χώρα για τον κύριο Σακασβίλη. Ξέρετε. Καλή παρατήρηση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το Λουξεμβούριο δεν έχει να πάρει μαθήματα για το πώς να προχωρήσει στην Προεδρία του. Τα ξέρετε πολύ καλά, είσαστε μια χώρα με εμπειρία από αυτού. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Να ηγηθείτε με πυγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το εξάμεινο αυτό με όραμα και στρατηγική. Η πρώτη μου παρατήρηση, το πρώτο μου σχόλιο είναι για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το TTIP, την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές ομάδες στηρίζουν τις διαπραγματεύσεις και θέλουν να καταλήξουν διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή. Αλλά Πέρα από το TTIP υπάρχουν άλλα σχέδια για να ενισχυθούν οι διατλαντικοί δεσμοί, οι δεσμοί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια κρίσιμη στιγμή σήμερα όπου θα έπρεπε να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο αυτών δυτικών συμμάχων. Δεύτερον, είπα τους εκπρόσωπος Μογκερίνη αναφέρθηκε σε στρατηγική όσον αφορά την ε, προπαγάνδα και θα ήθελα η κυρία Μογκερίνη πρώτα απ' όλα να φροντίσει για τη διοικητική ικανότητα αλλά και για την καλή κατανόηση του θέματος αυτού. Το έγγραφο πάντως που εγκρίθηκε αναφέρεται στην Ανατολική Γετνίαση. Εγώ καταλαβαίνω ότι η προπαγάνδα είναι ένα πολιτικό εργαλείο, ένα εργαλείο για πολιτικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσική Ομοσπονδία κυρίως προς τις δυτικές κοινωνίες. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα, όχι μόνο πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, αλλά πώς θα βοηθήσουμε και τις δικές μας τις χώρες, γιατί μπορεί να είμαστε τα αόρατα θύματα αυτής της προπαγάνδας. Θέλω λοιπόν να σχολιάσετε πάνω σε αυτό για την ε, πιο στενή συνεργασία και για το τι δράσεις πιστεύετε με δική σας πρωτοβουλία θα έπρεπε να αναλυφθούν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω με την τελευταία ερώτηση. Πρέπει να περιοριστώ έτσι κι αλλιώς. Το καταλαβαίνετε, πρέπει να πάω στη Γουιάννα. Και το αεροπλάνο φεύγει από τις Βρυξέλλες. Αν το χάσω, ε, δεν θα ε, μπορέσω να εκπροσωπήσω τη Φρεντερίκα Μογκερίνη στο Καρικόμ, στη Γουιάννα. Οπότε λυπάμαι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για το TTIP. Χτες ήμουνα στην Επιτροπή Ίντα και επί δύο ώρες συζητούσαμε για το TTIP. Ρωτάτε τη γνώμη μου. Ε, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επίμαχο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα, κατά τη γνώμη μου, θα εξαρτηθούν λοιπόν από το κατά πόσο θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια νέα γενιά μηχανισμού διαιτησίας, επίλυξης διαφορών, που να πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχω εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα υπάρχει TTIP, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Επιτροπή κάνει τις διαπραγματεύσεις κυρίως. Σίγουρα και η άποψη του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντική, αλλά εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε λόγο που βαραίνει όλος ιδιαίτερος στην απόφαση για τον ΕΙΤΟ στο τέλος. Και μπορούμε να παραλύσουμε την κατάσταση και με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ομπάμα είχε το Trade Promotional Authority το Κογκρέσο μπορεί να πει ναι ή όχι. Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είμαι σίγουρος Εννέα επιτροπές σας έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα μέχρι τώρα. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα βρουν τη σωστή λύση. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, επιτρέψτε μου να σας πω. Και το είπε στην αρχή και ο πρόεδρο. Υπήρξε χτες αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι ένα παράδειγμα αυτό που είναι σπάνιο τον τελευταίο καιρό. Α, Αμερικανοί, Ρώσοι, Ευρωπαίοι, τώρα με το Ιράν, όλοι μαζί κατάφεραν μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεις να φτάσουν σε μια πολύ σημαντική συμφωνία για την ειρήνη στον κόσμο. Όσον αφορά τώρα την Ουκρανία το Σακασβίλη. Νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει ο πρόεδρος. Στην Τυφλίδα μπορεί να υπάρχουν δισταγμοί, το ίδιο και στην Ουκρανία. Εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ στην εσωτερική πολιτική της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο την πήρε την απόφαση. Πάντως εύχομαι όχι μόνο στην ε, Οδυσσό στην Ουκρανία, αλλά και στις άλλες περιοχές καλή τύχη. Για τη Στρεμπρένιτσα τώρα, η Βοσνία. Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι είδα τις εικόνες και συναντήθηκα, όπως και άλλοι υπουργοί εξωτερικών, με τον ε, Βούτσιτς εδώ στις Βρυξέλλες. Mm. Είναι κάποιος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πού θέλει να πάει, προς ποια κατεύθυνση. Η συμπεριφορά του κατά κάποιο τρόπο ε, πώς να πούμε, παραδειγματική γιατί δεν απάντησε στις προκλήσεις. Η πρόσκληση τώρα που έγινε από τον Πρωθυπουργό Βούτσιτ στην Προεδρία της Βοσνίας Αρζεχοβίνης, να συναντηθούν στο Βελιγράδι, ίσως είναι ένα δυνατό μήνυμα. Και εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε κάποια μέρα να κάνουμε αυτό που αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη το 2003. Χωρίς τη Σερβία δεν γίνεται. Βέβαια και η Σερβία από την πλευρά της πρέπει να κάνει προσπάθειες και να συνεχίσει και αυτή τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους στην Πρίστινα είναι πολύ σημαντικό και είναι αποφασιστική σημασία, θα έλεγα, για τον δρόμο της Σερβίας προς την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα το Κωσυφοπαίδιο και την Κύπρο που με ρωτήσατε για το Κωσυφοπαίδιο, η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Συνεχίζονται οι εργασίες και ελπίζω πολύ σύντομα να περάσουμε στην υπογραφή, ελπίζω, πόλου Λουξεμβουργιανής Προεδρίας για την Κύπρο. προσλήθηκα ως Προεδρία να επισκεφθώ την Κύπρο. Θα συζητήσω λοιπόν. Κύπρος πιο στο νότο, Κύπρος πιο στο βορρά. Θα κοιτάξω λοιπόν με μηνύματα σαφή που ενθαρρύνουν και τις δύο πλευρές να προχωρήσω και να βοηθήσω να προχωρήσει η εξέλιξη θετική αυτή την εποχή. Στην προηγούμενη προεδρία μας πριν από 10 χρόνια ήμασταν και τότε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Πέρασαν 10 χρόνια όμως χωρίς συμφωνία. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν ήρθε τώρα η στιγμή με την βούληση και των δύο πλευρών στην Κύπρο και με την Προεδρία της Κύπρου και τους ομολόγους της στο Βορρά να καταλήξουν σε μια δυναμική που θα φέρει πιο θετικά αποτελέσματα. Για την Ουκρανία πάλι, ναι. Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε τώρα για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία κατά της διαφθοράς, αν μιλήσουμε για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή υφίσταται και μια εμπόλεμη κατάσταση σε ένα σημαντικό κομμάτι της επικράτειάς της. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε το κοινοβούλιο πάνω απ' όλα στο Κίεβο, αλλά και τις διάφορες πολιτικές αρχές να προχωρήσουν. Γιατί αν οι αρχές του Κιέβου οι Ουκρανικές αρχές δεν το κάνουν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η Ευρώπη εκείνη που θα το κάνει, με ό,τι βοήθεια και αν προσφέρει, δεν είναι η Ευρώπη που θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται λοιπόν θάρρος για να τις κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Εγώ δεν έχω πάντως τελευταία νέα από την Ουκρανία. Ξέρω ότι όταν πήγα στο Κίεβο υπήρξε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι επ' αυτού η διεθνής βοήθεια είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα να βγει από την τρύπα στην οποία έχει βρεθεί. Από την άλλη μεριά, αν θέλουμε να σταθεροποιηθεί η Ουκρανία, αυτό δεν θα γίνει δωρεάν. Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να κάνουν προσπάθειες. Όσον αφορά τώρα το μας, βλέπω κάποιους συναδέρφους και υπουργού Εξωτερικών και την κυρία Φωτίγκα, διάφορους εδώ μεταξύ σας και πραγματικά χαίρομαι πολύ για την έρευνα που ρωτήσατε. Ξέρω ότι τη Δευτέρα ο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων των Κάτω Χωρών πήγε στη Νέα Υόρκη. Και εγώ πήγα στο Σεβούλιο Ασφαλείας πριν από ένα χρόνο και συζητήσαμε είναι μια έρευνα η οποία γίνεται από έναν ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό. Ο Διεθνής Οργανισμός Αεροπλοίας, αν αναπατώμε. Αυτός το έχει αναλάβει για την πτήση αυτή των μαλισιανών αεροπορικών γραμμών. Τώρα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να πείτε οτιδήποτε. Ελπίζω να βρεθούν υπεύθυνοι, να φανεί ποιο φταίει. Αλλά δεν θέλω να κάνω πως ξέρω ποιος φταίει για αυτό το φοβερό δράμα. Ελπίζω κι εγώ, όπως όλοι οι πολίτες, ότι κάποια μέρα η αλήθεια θα λάμψει και οι θεσμοί, τα όργανα που δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα θα καταλήξουν. Τώρα η συζήτηση κατά τα άλλα έχει γίνει πολλές φορές. Δεν έχουμε καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι υπηρεσίε οι εξωτερικές πρέπει να μπορούν να έχουν βοήθεια από τα προξενία σε όλες τις χώρες κόσμου. Υπάρχουν ακόμα κάποια εμπόδια. Δεν ξέρω αν θα τα ξεπεράσουμε κάποια μέρα, πάντως είναι θέμα ανατροπίας. Πιστεύω πως αν μιλάμε για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, πρέπει από την άλλη μεριά να μιλάμε και ευρωπαϊκά όργανα και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι ευρωπαϊκή και τα προξενία θα έπρεπε να μπορούν να βοηθούν όλους τους Ευρωπαίους άπαξ και έχουν κάποια ζητήματα επίγοντα και προσφεύγουν στα προξενία. Ένα ακόμα πράγμα μένει να σας απαντήσω. Ναι, η Άννα Φωτίγκα. Ρώτησε το εξή. Για τη Σερβία. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εσωτερικών στο Συμβούλιο Τσάι, Εσωτερικών Υποθέσεων και δικαιοσύνη και είπα, και νομίζω ότι το ξέρει και αυτός όπως και ο υπουργό Εξωτερικών, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με την διεθνή πολιτική. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί δηλαδή περισσότερο σε αυτές τις θέσεις. Είναι σημαντικό. Η Σερβία προς το παρόν τηρεί 60% μόνο των θέσεων που έχουν υιοθετηθεί. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να βελτιωθεί. Και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό πολύ σοβαρά. Όσον αφορά λοιπόν... Α, ναι, Έντουαρτ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου. Και πράγματι, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στα Βαλκάνια, υπάρχουν και θετικά. Ο διάλογος ανάμεσα στην Πριστίνα και το Βελιγράδι μπορεί να καταλήξει όχι αμέσως, αλλά να καταλήξει θετικά. Η πρωτοβουλία αυτή στη Βοσνία Ζεγοβίνη που ανελήφθη από τους Γερμανούς και τους Άγγλους και τώρα είναι υπό την αρμοδιότητα τη Σοντερίκα Μογκερίνη, μπορεί να βοηθήσει προ τη σωστή κατεύθυνση. Οι άνθρωποι στη Βοσνία Αζεκοβίνη βέβαια πρέπει να δεχτούν ότι ζουν σε μία χώρα και όχι ότι πρόκειται για δύο-τρία έθνη που ζουν το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Η συνάντηση στο Σαράγεβο που θα γίνει θα μας βοηθήσει πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, για την τέως γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπράβο για το έργο σας. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ και τον Επίτροπο Χάν, διότι ήταν δύσκολο. Πέντε μέρες είπατε ότι διαπραγματευόσασταν. Το πρόβλημα εκεί είναι, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, βρήκαμε έναν τρόπο να μιλήσουμε με τους Έλληνες. Γιατί βλέπετε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υποψήφια μια χώρα και μετά για δέκα χρόνια να μην αλλάξει τίποτα. Δεν έχει νόημα. Δεν λέω ότι φταίει η Ελλάδα. Δεν το λέω αυτό. Δεν είναι δικιά μου υπόθεση αυτό. Αλλά τώρα η Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση. Ελπίζω να βελτιωθεί περισσότερο η κατάσταση στο μέλλον και γίνεται αυτή η προσπάθεια στη χώρα, στα Σκόπια. Ελπίζω να βρεθεί μια καλή συνεργασία και να βρεθούν και καλές λύσεις και να μην μείνει η χώρα αυτή έτσι. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την κατάσταση. Δεν φταίει η Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη μπορούσε να είναι πιο κοντά και να αναμειγνώταν περισσότερο στο κράτος δικαίου της χώρας αυτής, ίσως να είχαμε μπορέσει πιο γρήγορα να διορθώσουμε την κατάσταση. Πάντως, καλή τύχη στην πρωτοβουλία σας. Είναι θετική. Ευχαριστούμε πολύ, Ζω, για την παρουσίασή σου. Καλό ταξίδι και θα χαρούμε πάρα πολύ να σε ξαναδούμε. Ερχόμαστε τώρα. Το επόμενο σημείο, ποιο είναι το επόμενο σημείο? Συμφωνία πλαίσιο συνολική εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη και του, της Δημοκρατίας του Βιετνάμ. Είναι η Μπάρμπαρα Λοχμπιλτερ η οποία είναι συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει για αυτήν την ε, συμφωνία εταιρικού χαρακτήρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ και αυτή είναι το επιστέγασμα μιας, ε, συμφωνία, μιας διαδικασίας 25 ετών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Θα είχε ε, εγκριθεί ήδη αυτή η συμφωνία πριν από τρία χρόνια, αλλά δεν υπήρχε η θετική γνώμη όλων των κοινοβουλίων. Το Βιετνάμ έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες κύρωσης ήδη από τον Νοέμβριο του 2013. Αυτό το οποίο χρειάζεται από την ευρωπαϊκή πλευρά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι χρειάστηκαμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για την κύρωση και αυτό δεν το καταλαβαίνει η εταίρα χώρη μας. Ίσως θα πρέπει το θέμα αυτό να συζητηθεί και με την κυρία Μογκερίνη στα πλαίσια της ε, συζήτησης για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ε, ασφάλειας. Η συμφωνία με το Βιετνάμ λοιπόν είναι το, η συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μας με το Βιετνάμ. Από το 2012 υπήρξαν συζητήσεις επίσης για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου όπου ε, εργάζονται οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΣΥΝΤΕ. Επίσης υπάρχει και μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο άρθρο 1 και το άρθρο 57 επίσης αναφέρει ότι σε περίπτωση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ανασταλεί η εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η η συμφωνία θα δημιουργήσει μια νομική ρήτρα ώστε να υπάρχει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσω της συμφωνίας αυτής ανθρωπίνων ε, ελευθερών εμπορίου. Και πιστεύω ότι η Κομισιόν μπορεί να το επιβεβαίωσει αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε μια θετική γνώμη για αυτή την έκθεση. Θα ψηφίσουμε απλώ ναι ή όχι. Και εγώ ως εισηγήτρια προφανώς θέλω να σας προτείνω να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή έχει λεπτομεριακές πρόνοιες για τις μελλοντικέ σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ. Το σχέδιο ε, έκθεσης έχει βέβαια συγκεκριμένες ε, μορφές περιορισμού σε σχέση με, την, ε, με το μήκος της έκθεσης αυτής και χρειάζεται να περικόψω στο ίμιση την αρχική μου έκθεση. Είναι πολλά θέματα λοιπόν τα οποία για το λόγο αυτό δεν μπόρεσα να τα διαλάβω. Ελπίζω λοιπόν ότι οι συνεισηγητές θα μπορέσουν να συμπληρώσουν όλα αυτά με τις τροπολογίες τους. Το Βιετνάμ έχει κάνει τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των στόχων της χιλιετίας. Μείωση της ένδυας, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική προστασία δημιουργία θέσεων απασχόληση και υγειονομική περίθαλψη. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ επίσης γνωρίζει πολύ καλά ότι η πολιτική ντόιμόη, η πολιτική ανανέωσης έχει οδηγήσει και σε αρνητικά αποτελέσματα. Έχει υπάρξει μεγαλύτερη ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματο, χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, καταστροφή του περιβάλλοντο και εδώ είναι απαραίτητε νομοθετικέ από απαραίτητε για να αντιμετωπιστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος και η αποψήλωση των δασών. Η διαφθορά είναι και ένα τμήμα του προβλήματος. Η έκθεση επίσης αναφέρεται και στην απαλωτρίωση γεών και άλλων ιδιοκτησιών από τις αρχές του ε, Βιετνάμ. Υπάρχει και μία περιστολή των πολιτικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου. Βάσει του δίκτυ για την ε, ελευθερία του τύπου από 180 χώρες στο Βιετνάμ βρίσκεται στη θέση 175, απαγορεύεται τα ανεξάρτητα συνδικάτα και υπάρχουν ε, περίπου 650 άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Λόγω της ε, έκτασης των ανθρωπίνων, της παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η Κομισιόν να ακολουθήσει την ε, θέση της ε, διαμεσολαβήτριας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρξει μια μελέτη ώστε μάλλον να αναφερθεί και στην ε, συμφωνία αυτή πλήρως στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει όλα αυτά να μας προωθήσουν σε ένα συγκεκριμένο διάλογο, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να οδηγήσει σε πραγματική πρόοδο για την επιβολή ενός κράτους δικαίου και για την διατήρηση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Βιετνάμ είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του, των ΗΕ αυτή τη στιγμή και επομένως έχει κάθε συμφέρον αυτά τα οποία του ζητούν οι περιοδικές εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα εφαρμόσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες βελτιώσεις στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες προβλέπονται τώρα να γίνουν από την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στην βελτίωση της κατάστασης με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού υποβολής ε, παραπώνων από άτομα και ενώσεις όταν μέσα στα προγράμματα, μέσα από τα προγράμματα των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύονται οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή προκαλούνται τέτοιες δια, ε, παραβιάσεις. Επίσης είναι σημαντικό να γίνουν όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορέσουν να απαλληλθούν οι εντάσεις στη, στο νότιο κινέζικο πέλαγος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και περιμένω και τα σχόλια των συνεισηγητών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όμως και την κυρία Λόχμπιλερ για την έκθεσή της. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την κύρωση αυτής τη συμφωνίας πλαίσιο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν οι αντισυμβαλόμενοι να Είναι σφαιρική συμφωνία που καθορίζει αλλά και διευρύνει τις σχέσεις μας με την δημοκρατία του Βιετνάμ και καλύπτει οικονομία, εμπόριο, επενδύσεις αλλά και ενέργεια όπως και συμφωνία σε θέματα συνεργασία, θέματα ασφαλεία. Να δούμε τώρα κάποια επιμέρου στοιχεία αυτή τη εταιρική σχέση. Πρώτα-πρώτα ότι χρειάζεται να υλοποιηθούν κάποιε μεταρρυθμίσει όπω τα λέει πολύ σωστά η κυρία Λόχομπλη στο κείμενο. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο τη συμφωνία θα πρέπει να γίνουν σεβαστή η αρχή τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πολύ βασικό. Δεν θα πρέπει κανεί να λησμονεί ότι παρά τη σχετική οικονομική επιτυχία της χώρας βασικά εκεί πέρα υπάρχει μονοπόλιο. Υπάρχει μονοκομματικό καθεστώς και δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Άρα κάπως ρίψω ε, κίνδυνο να θεωρεί ότι εκεί πριν ανέβει η δημοκρατία. Ε, έχουμε την καταστολή των ε, κομμουνιστών, αλλά βέβαια πάρα πολλές ε, μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει όσον αφορά την δικαιοσύνη, αλλά και διώξεις μειονοτήτων τους, τους λόφους, τους, τους χριστιανούς και άλλους. Και κύριε Λόχμπιλερ το ανέφερε Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέτρα έχουμε στην διάθεσή μας με ρεαλιστικό τρόπο. Πέραν αυτών πάντως οι σχέσεις με το Βιετνάμ ανάγονται στην τελευταία 25 ετία οπότε αυτή η συνεργασία εταιρική σχέση και συνεργασίας ωφελεί και, τους, και τα δύο μέρη κυρίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και με αυτή τη συμφωνία αλλά και συμφωνία ε, ελευθέρων συναλλαγών που τώρα την πραγματευόμαστε θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε τώρα πρόσβαση σε μια πολύ δυναμική αγορά όπου ο πληθυσμός όλο ένα αυξάνει. Είναι εντυπωσιακό ο δυναμικός ρυθμός της εξέλιξης ε, του πληθυσμού. Επίσης η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για ξένες επενδύσεις. Οπότε πάνω σε αυτό θα συνεργαστούμε. Οπότε αυτή η εταιρική σχέση και οι ελεύθερες συναλλαγές θα είναι κάτι βασικό για τη σχέση μας με ναι, την ευρύτερη περιοχή του ΑΣΕΑΝ. Αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται θαλασσία ασφάλεια, τρομοκρατία και την κυβέρνηση ασφάλεια. Η χώρα δραματίζει σημαντικό ρόλο εκεί στην περιφέρεια ιδίω όσον αφορά τι διαφορέ για την νότια θάλασσα τη Κίνα ε, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με κάποιε σοβαρέ απειλέ που υπάρχουν εκεί και είναι κίνδυνο για το εμπόριο. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια συμφωνία με τη βάση του εθνού δικαίου. Πάντως υπάρχουν κάποιε απειλέ από την Κίνα και έχει γίνει κάποια προσέγγιση με τι ε, ΗΠΑ και τους άλλους ε, ε, εταίρους τη περιοχή για να ανασχέσει αυτή την επιθετικότητα από την Κίνα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ρώσιμο το 2016 που θα στην αυτή η συμφωνία. Θα είναι μεγάλο βήμα για το μέλλον της χώρας. Από πολλές απόψεις βέβαια ακόμα θα πρέπει να δούμε τι λύση θα δώσουμε. Και επομένως τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την επιρροή της στην Ασία και να βοηθήσει για να πρετανεύσει η ειρήνη, κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η ασφάλεια κατά θάλασσα. Επομένω, καταλήγοντα, πρέπει να σα πω ότι θεωρώ παρακολουθητική αυτή την ε, έκθεση και είναι πολύ θετικό το πώς συνεργαστήκαμε με τους άλλους ε, εισηγητές και την ε, κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριος Μπετίνη. Εγώ συμφωνώ. Επομένως με, με τη γενικό πνεύμα της έκθεσης Φεύγω και θεωρώ θετική αυτή τη συμφωνία, μια που το Βιετνάμ είναι μια περίπλοκη χώρα. Έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου στον οικονομικό τομέα, αλλά επίσης και από πλευράς πολιτιστικής. Να μην ξεχνούμε ότι το παρελθόν της χώρας ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δραματικό. Οπότε με αυτά τα βήματα προόδου ε, πετύχανε να θεσπίσουν ένα νέο σύνταγμα. Βέβαια, πάρα πολλέ φορέ παραμένουν τα συντάγματα νεκρό γράμμα. Αυτό το ξέρουμε από την ιστορία και την ευρωπαϊκή ιστορία. Παρ' όλα αυτά, από όσο αντιλαμβάνομαι, οι ηγέτες της χώρας προσπαθούν να υλοποιήσουν τις βασικότερες αρχές. Ακόμα βέβαια σοβούν σημαντικά προβλήματα. Επίσης η υλοποίηση αυτών που έχουν υποσχεθεί θα κάνουν κατόπιν κάποιες συστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκής κοινότητας. Και κάθε φορά που συναντούμε κάποιες συμφωνίες, ακόμα και εμπορικές, πολλές φορές όταν αφορούν κάποιες χώρες όπου ακόμα δεν είναι αυτονόητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές ελευθερίες θα πρέπει τους βασικούς μας στόχους εκεί να τους ε, προωθούμε. Και θα πρέπει κάπως να τίθενται κάποιες προθεσμίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση αυτών των αρχών. Οπότε θεωρώ ότι και με αυτή μας την έκθεση θα πρέπει να προωθούμε αυτές τις αρχές, να πιέζουμε το ώστε να υλοποιηθούν ε, αυτές οι συστάσεις. Ακριβώς αυτό το οποίο κάνει η συνάδελφος Λόχμπιλερ. Άρα θα πρέπει εκεί να βρούμε την σωστή ισορροπία και η ισορροπία δεν εννοώ ότι θα πρέπει κάποια από αυτά τα θέματα να τα υποτιμήσουν αλλά θα πρέπει όλες τις χώρες με τις οποίες κάνουμε συμφωνίες να τις μεταχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί για τελευταίου τελευταίο μήνες και εβδομάδες ασχολούμεθα με το τι θα γίνει με την Κίνα, με τη, κάποιες συμφωνίες ε, ε, εμπορικές. Επίσης έχουμε ασχοληθεί και με συμφωνίες εμπορικές με το Τουρκμενιστάν αλλά τι γίνεται εκεί με το περιβάλλον, τι γίνεται με το εργατικό δίκαιο και τα ανθρώπινα μέσα στις χώρες εκείνες. Νομίζω εκεί τα πράγματα είναι αρκετά στριμωγμένα, περίπλοκα και δεν νομίζω ότι η ηγέτες των χωρών αυτών λαμβάνει υπόψη αυτές τις αρχές. Όλα αυτά όμως προχωρούμε και ολοκληρώνουμε τη συνέψη κάποιων συνθήκων. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο ισόρροπο, ισορροπημένο, δίκαιο να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις χώρες. Να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά δηλαδή. Uh, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Μας δίνει ένα συνολικό πλαίσιο για τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το Βιετνάμ. Είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο του παγκόσμιου εμπορικού στερεώματος, αλλά φαίνεται ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση υπολείπεται πολύ από την εφαρμογή των απαραίτητων κοινωνικών μεταμορφ... Ε, μεταρρυθμίσεων. Είναι πολλές οι εθνοτικές μειονότητες οι οποίες παραμελούνται ή αγνοούνται τελείως από την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο αλφαβητισμού ή σχολικής προσέλευσης στο Βιετνάμ. Υπάρχουν ε, εκθέσεις για καταστολή μειωτικών γλωσσών και αρπαγής γης. Με το Κομμουνιστικό Σύνταγμα του Βιετνάμ όλη η γη ανήκει στο κράτος. υπάρχουν επίσης θέματα ελευθερίας του τύπου ενδημική διαφθορά των αξιωματούχων του κόμματος σε όλα τα επίπεδα. Αλλά παρά το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρξει πίεση προ την κυβέρνηση του Βιετνάμ για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίσει την εφαρμογή και την εφαρμογή μια φιλόδοξή συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να έρθει από μέσα και όχι από του διαδρόμου των Βρυξελών. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με το Βιετνάμ λοιπόν θα δώσει πολύ περισσότερες δυνατότητε να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία οι πολίτες του Βιετνάμ και να βγουν μέσω του εμπορίου από την ένδια. Μια τέτοια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα οδηγήσει και σε σταθερότητα και προβλεψιμότητα που είναι απαραίτητη για τους επενδυτές μας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει ισότης ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών εταιριών για να αντιμετωπίσουμε τα εμπορικά μας συμφέροντα από τα οποία εξαρτώνται τόσες πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη να υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος των κανόνων προέλευσης. Ελπίζω λοιπόν ότι και αυτή η συμφωνία και η ιατρική σχέση και η συμφωνία ελευθερών εμπορίου θα φέρουν ευμάρια και στο Βιετνάμ και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την συγκίτρια για το σχέδιο έκθεσης. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί έχουμε το θέμα αυτό ενώπιόν μας. Αν λάβουμε υπόψη την αυξανόμενη σημασία της ε, βελτίωσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ, εγώ υποστηρίζω απόλυτα το να υπάρξει συμφωνία για τα θέματα αυτά. Για το Βιετνάμ πιστεύω ότι η ενίσχυση των σχέσεων του με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη προτεραιότητα τη στιγμή που αντιμετωπίζει πολύ σημαντικέ προκλήσει και οικονομικά αλλά και πολιτικά. Η ένδια έχει μειωθεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ανισότητα και είναι μεγάλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό που αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο το χρόνο μια συνολική συζήτηση θα έχει μεγάλη σημασία για τις ε, εξαγωγές του Βιετνάμ που αυξάνονται προς το παρόν σε επίπεδο μόνο 5,4% το χρόνο. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε αυτήν την περιοχή του κόσμου μετά από το τέλος της ασιατικής κρίσης. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρος στο Βιετνάμ, στην Ασία και είναι σαφές ότι για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασιατικών χωρών οι εταιρικές αυτές σχέσεις έχουν ενισχύσει πολύ τη συνεργασία και έχουν στρατηγική σημασία. Κάποιες παρατηρήσεις μοναχα για το σχέδιο έκθεση και εγώ υποστηρίζω τους φιλόδοξους στόχους που θέτει η εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να έχουμε μια σαφή προσέγγιση για το πού θέλουμε να φτάσουμε στα επόμενα πέντε χρόνια σύγχρονο όμω. θα πρέπει να δούμε πώ υποστηρίζουμε το Βιετνάμ για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ευκυβερνησία. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μόνο αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και τα πρότυπα τα οποία επιζητούμε. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν μεγαλύτερη έμφαση στο σημείο αυτό και χαιρετίζω την παράγραφο 4 για την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη ικανότητα του Βιετνάμ για το κράτος δικαίου και την καλή δημόσια διοίκηση. Στην παράγραφο 21 επίσης υποστηρίζω το να εστιάσουμε, να δώσουμε μια έμφαση στην ανάπτυξη βιώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης θα πρέπει να εστιάσουμε και στο γεγονός ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα διαφθοράς, ανισότητας των φύλων, προστασίας του περιβάλλοντος αν αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μέσω της συμφωνίας υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση ώστε το Βιετνάμ να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Πρέπει ιδιαίτερα να εξασφαλίσουμε ότι θα τους δώσουμε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και όχι απλώς να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό αναπτυξιακής βοήθειας κατά 30% όπως λέγεται εδώ. Πρέπει να πράξουμε περισσότερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων <clears throat> και της ανάπτυξης και το θέμα των βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης είναι επίσης σημαντικό. Ενώ το κάνουμε αυτό, η Κομισιόν να εξετάσει την ε, ορατότητα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βιετνάμ. Ξέρω ότι είμαστε σε ανταγωνισμό με άλλες πολλές χώρες και οντότητες. Ίσως η Κομισιόν θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα για το πού χρηματοδοτούμε. Εγώ υποστηρίζω αυτά που είπε η συγκήτρια να υπάρξει μια νομική σύνδεση μεταξύ τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και να υπάρχει δυνατότητα αναστολή τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου αν υπάρξουν σοβαρέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ζητάει η συγκήτρια επίση να υπάρξει μια <clears throat> έκθεση αντικτύπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Συμφωνία ε, του Ελευθέρου Εμπορίου, όπω ζήτησε και η διαμεσολαβήτρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα όμως να ρωτήσω την Κομισιόν τι έγινε με την γνωμοδότηση που θα δημοσίευε η κυρία Μάλουσον για το θέμα αυτό μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δεν είναι σαφές πότε τώρα θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτή η έκθεση. Ξέρω ότι δεν είναι ένα δημόσιο έγγραφο. Θα ήταν χρήσιμο εμείς ως βουλευτές να έχουμε αυτές τις πληροφορίες στα χέρια μας. Και τέλος θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό το θέμα της εμπορίας ανθρώπων και άλλοι συνάδελφοι το έχουν θίξει, αλλά είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι μια από τις χώρες που έχουμε το μεγαλύτερο βαθμό εμπορίας ανθρώπων και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση αυτή τη μάστιγος και να έχουμε μια συντονισμένη αντιμετώπιση από τα κάτι μελη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ προ, προσβλέπω σε συνεργασία με την εισηγήτρια πρωτού φτάσουμε στο τελικό στάδιο τη έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλντερ. Μπορείτε να είστε σύντομοι για να μας πληροφορήσουν ο κύριος Κούκαν και ο κύριος Χάουιτ για τα γεγονότα στα Σκόπια. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κύριους συζητητές για τις, ε, τα σχόλιά τους και όπως είπα και στην αρχή πρέπει η έκθεσή μου να είναι σύντομη. Όλα τα θέματα που έχετε αναφέρει είναι πολύ χρήσιμο αν μπορείτε να τα μετατρέψετε σε τροπολογίες Ιδίω για το θέμα που ανέφερε η κυρία Γκίλ, το θέμα της εμπορίας ανθρώπων, είναι κάτι που είναι σημαντικό να παραπέμψουμε και στην πρωτοβουλία των χωρών ΑΣΕΑΝ να υπάρξει μια ανεξάρτητη σύμβαση για τα θέματα εμπορίας ανθρώπων, όπου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το Βιετνάμ. Ευχαριστώ. Πού είναι ο κύριος Κούκαν? When we start then it's over. Μα τότε δεν μπορούμε να το κάνουμε, λέει ο πρόεδρος Μπροκ. Excuse me. Ε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μήπως θα μπορούσατε να ζητήσετε από την Επιτροπή να επανέλθει. Πολύ καλή ιδέα, λέει ο πρόεδρος. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, εδώ εκπροσωπώ τη Γενική μου Διεύθυνση σήμερα και επειδή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τις διμερείς ε, συνομιλίες ε, για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, δια συνάδελφοί μου τώρα είναι στο ανώ για τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών και μετά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια πολιτική απόφαση για το πώς θα πρέπει να είναι η πολιτική συμφωνία. Σημείωσα όλα τα σχόλια το, της εισηγήτριας και των άλλων ομιλητών. Ξέρετε, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω 100% ότι για το ποιο θα είναι το περιεχόμενο στη συμφωνία αυτή. Όμως πιστεύω ότι θα προβλέπονται διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα ή έμεσα με την βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μπορώ ήδη να σας πω ότι αυτά που βάζουμε στις διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους μας από το Βιετνάμ είναι να αναφέρεται σαφώς το προήμιο η αρχή του FTA, της ε, Μπορικής ε, Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο είναι το εξή. Άκουσα ότι θέλετε μια σύνδεση νομική και θεσμική ανάμεσα στο FTA και το PCA, ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ρήτρε μη εκτέλεσης που επιτρέπουν βασικά να υιοθετήσουμε μέτρα για την πάυση του PCA και ενδεχομένως και του FTA. Αυτά τα βάλαμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει τέτοια σύνδεση θεσμική ανάμεσα στο FTA και το PCA. Τώρα για τον μηχανισμό των ανεξάρτητων ε, προσφυγών. Υπάρχουν διάφορες ε, διατάξεις από αυτού και στα διάφορα κεφάλαια αλλά και σε όλα τα θεσμικά οι διατάξεις του FTA που μιλούν για ειδικά όργανα, εμπορική επιτροπή, SPS ή οτιδήποτε άλλο για τα διάφορα κεφάλαια τα προβλέπονται διατάξεις που θα επιτρέπουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γύρουν τις ανησυχίες τους και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ισχύει και για το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξης, όπου υπάρχει μια εσωτερική ομάδα συμβουλευτική, δύο μάλλον τέτοιες, μία στο Βιετνάμ και μία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μέσω αυτού του μηχανισμού οι διάφορες κοινότητες ενδιαφερόμενοι μπορούν να γύρουν ε, παράπονα άπαξ και πιστεύουν ότι έχουν θέση. Υπάρχει και κεφάλαιο στην συμφωνία στο FTA για τη διαφάνεια. Υπάρχουν διατάξεις που λένε ότι υπάρχει το δικαίωμα σχολιασμού και οι πλευρές του FTA πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτά τα σχόλια. Αν δηλαδή υπάρχει μια νομοθεσία ή κάποιο νομοθετικό πλαίσιο οι ενδιαφερόμενες πλευρές μπορούν να υποβάλουν σχόλια και οι αρχές είναι υποχρεωμένες να τα λάβουν υπόψη τους τα σχόλια αυτά. Και αν δεν γίνει αυτό και μια πλευρά έχει λόγο ένστασης, υπάρχει ο μηχανισμός που μπορούν να τεθούν αυτές οι ενστάσεις και υπάρχει και το δικαίωμα της αναθεώρησης και προσφυγής αυτών των μέτρων και το δικαίωμα σε απόφαση βάσει αποδείξεων και πρακτικών. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο για τη διαφάνεια του FTA τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά, συμπεριλαμβάνει αυτές τις διατάξεις. Αυτά αναφέρει το PCA. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία μέσα από τα οποία προσπαθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα βάλουμε στο κέντρο των σχέσεών μας με το Βιετνάμ. Ξέρω ότι η κυρία Λόχ Μπίλερ στις 12 Μαΐου συμμετείχε σε μια εκδήλωση που οργανώσαμε με τους συναδέλφους μας από το ΔΙΕΣ αλλά και από άλλες γενικές διευθύνσει. Η εκδήλωση αυτή ήταν αφιερωμένη στο πώς αντιμετωπίσουμε το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διμερείς μας σχέσεις με το Βιετνάμ. Έχουμε και ένα εγγραφό που συμπεριλαμβάνει συνοπτικά όλες τις συστάσεις που έγιναν από εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων στην εκδήλωση αυτή. Υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ήδη στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Και τώρα συντάσσουμε έκθεση στην οποία εξηγούμε ότι εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, λέμε ποιες διατάξεις στο FTA, στη συμφωνία αυτή δηλαδή, αναφέρονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, πώς πρέπει να ερμηνευτούν και πώς θα τεθούν σε εφαρμογή. Και αυτό με, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν ή θα αναπτύξουμε. Οι συνάδελφοι τώρα από τις άλλες γενικές διευθύνσεις δεν είναι εδώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι για την αναπτυξιακή συνεργασία υπάρχουν πολλά χρήματα τα οποία πηγαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και την βιώσιμη ανάπτυξη. Και μέσω του ενισχυμένου διαλόγου που θα έχουμε μετά την εφαρμογή του FTA θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει καλύτερος συνδυασμό δυνάμεων ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια με τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν και οι ανησυχίες που υπάρχουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, επανέρχομαι λίγο στο θέμα της ε, μελέτης επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο θέμα για όλους μας. Θέλω να επιθυμίσω ότι ο Επίτροπος Μάλστρομ πρόσφατα όταν είχε πάει στην Επιτροπή Ίντα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι και το εμπόριο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προωθούμε βασικές μας αρχές, τις διμερείς μας σχέσεις. Από το 2011 και μετά λοιπόν έχουμε δεσμευτεί να συμπεριλαμβάνουμε την αξιολόγηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε είδους έκθεση αξιολόγησης που κάνουμε όσον αφορά διαπραγματεύσεις για εμπορικές σχέσεις. Το Βιετνάμ είναι μια δική περίπτωση βέβαια. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται και όπως είπε και η Επίτροπος Μάστρομ στις 12 ε, Μαΐου στην εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκα πριν, η Επιτροπή πιστεύει ότι θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα η συμφωνία. Δεν θα υπάρχει έκθεση αξιολόγηση τώρα, αλλά θα υπάρχει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ε, διαπραγματεύσεων, στην επόμενη αξιολόγηση δηλαδή, θα υπάρχει και αξιολόγηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Λίγα λεπτά μας έχουν μείνει μόνο. Ο κύριος ε, Κούκαν πρέπει να φύγει σε 15 λεπτά, αλλά πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να μας εξηγήσει για τη συμφωνία που πέτυχε τη νύχτα. Ο κύριος Κούκαν μπορεί να αρχίσει και μετά και οι υπόλοιποι. Α, ήρθε και ο κύριος Χόουιτ. Ποιος θα αρχίσει. Όχι, μην φεύγετε. Άρχιστε κύριε Κούκαν, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ το ένα ακόμα γύρω διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν πριν από αρκετούς μήνες. Πρώτα πρώτα είχαμε τρεις ευρωβουλευτές που συνάντησαν τους ομολόγους τους στους οποίους είχε δοθεί εντολή από το κόμμα του Γκρούευσκη και τον Ζόραν Ζάγεφ, τον ε, ηγέτη της αντιπολίτευσης. Στις 2 Ιουνίου υπεγράφει η συμφωνία από τους ηγέτες και των τεσσάρων πιο σημαντικών πολιτικών κομμάτων της Μακεδονίας. σε συνεννόηση με το κόμμα της ε, αντιπολίτευσης, με τον κύριο Γκρουεύσκη και με τον κύριο ε, ηγέτη της αντιπολίτευσης και επίσης ε, το κόμμα που του Αλβανού Αλβανούς στον συνασπισμό που κυβερνά. Και έτσι πέρασε αυτή η συμφωνία. Εκεί Καλύτερα το πιο σημαντικό που ζήτησε η αντιπολίτευση, δηλαδή πρόορες εκλογές. Συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν τέτοιες πρόορες εκλογές τον Απρίλιο του χρόνου. Και αυτό το οποίο δεν συμφωνήθηκε είναι το πώς θα οργανωθεί η κυβέρνηση, ούτως ώστε να προετοιμάσει τη χώρα εν ώψη των εκλογών. ακριβώ και αυτό ήταν το ζήτημα το οποίο χθε και σήμερα συζητήθηκε μέχρι το ξημέρωμα. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε στις λεπτομέρειες, αλλά πρόεδρε το πιο σημαντικό για το κυβερνόν κόμμα ήταν η παρέτηση του Πρωθυπουργού. παρέτηση επομένω του πρώτου κυβέρνηση και τη κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ε, μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία πρόκειται να ε, προλυάνει το έδαφο για τι εκλογέ. Κάτι με το πιο σημαντικό θέμα για την αντιπολίτευση και τον ηγέτη Ζάεφ ε, ήταν το να υπάρξει μια υπηρεσία με επικεφαλής στον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος θα διερευνήσει εκείνες τις παγιδεύσεις συνομιλιών, ε, μαγνητοφωνή συνομιλιών επομένως, όπου θα έπρεπε να αποδειχθεί η γνησιότητά τους. Και όχι το ότι είναι κάτι το φτιαχτό. Αυτά είναι τα πιο καθόδη ζητήματα τελικά. Πάντως, κατέστη δυνατόν να μπορέσουμε να βρούμε ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την επιστροφή της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Και είπαμε ότι θα δουν σε αντιπολίτευση ε, κάποιες θέσεις υπουργών ή μάλλον υφυπουργών για να συμμετάσχουν στην διαδικασία. Και επίση η πιο σημαντική θέση δηλαδή, του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι για την προπαρασκευή των εκλογών τόσο σημαντική, θα δοθεί στην αντιπολίτευση. Αλλά, αλλά, υπό την προπόθεση ότι θα ήταν κάποιο τεχνοκράτη, κάποιο που έχει επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά το σχετικό θεματολόγιο, τα θέματα δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό θα οριστεί από την αντιπολίτευση κατόπιν συνεννόησης με το κυβερνόν κόμμα όπου στο εσωτερικό θα έχει όλες τις αρμοδιότητες του σχετικού χαρτοφυλακίου. Τώρα, η τάρα Υπουργεία, η Υφυπουργεία, που θα είναι στην υπηρεσία κυβέρνηση, δηλαδή Υπουργείο Εργασία, Υπουργείο Οικονομικών. Ρίτσαρτ, ποιο άλλο είναι. Ε, το Υπουργείο Γεωργία, αλλά και Κοινωνική Προνοία, λέει ο κ. Χάουιτ. Αυτά Συνεχίζει ο κ. Κούκαν, πρόκειται να κρυθούν Όμως, όταν έρθει η ώρα να ορίσει η αντιπολίτευση τους υφυπουργούς, θα μπορεί το κυβερνόν κόμμα επίσης να ορίσει τους εκπροσώπους τους ή στο σχετικό Υπουργείο που θα έχουν και οι σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και οι κυρίες. Άρα θα υπάρξει κάποια δυστυχία με το τι θέση θα πάρει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, διότι η πρώτη σημαντική ημερομηνία είναι η 1η Σεπτεμβρίου, διότι τότε η αντιπολίτευση θα επιστρέψει στη Βουλή. Θα επιστρέψει ούτω ώστε να παρίσταται για όλα τα σημαντικά τα οποία θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν εκεί στο Κοινοβούλιο. Αλλιώ δεν είναι δυνατόν με απουσία τη να προετοιμαστούν οι εκλογές. Σας προείπα ότι για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την ε, τήρηση αυτής της συμφωνίας. Γιατί θα θυμάστε καλά, Πρόεδρε, και εσείς, επί Επιτρόπου Φίλε και με την συμβολή του κυρίου Μπούζεκ αλλά και του κυρίου Χάουιτ τότε είχαμε καταφέρει να αποστάσουμε συμφωνία των πολιτικών κομμάτων. Είχαν προσυπογράψει μια συμφωνία. Και έτσι είχε εξασφαλιστεί η, συμφωνία, η συμμετοχή της ε, αντιπολίτευσης στις εκλογές, αλλά από τότε δεν εφαρμόστηκε εκείνη η συμφωνία. Άρα δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια. Και ήταν πάρα πολύ κακό αυτό για τη χώρα. Τώρα με τη συμφωνία η Μακεδονία νομίζουμε θα έχει την ευκαιρία ούτως ώστε να προοδεύσει και να ξεκινήσει τη διαδρομή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το timing για τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει την έκθεση προόδου. επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει με την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ βρίσκονται στην αίθουσα αναμονή τόσο καιρό. Και νομίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία ούτως ώστε να δοθεί μια λύση στο θέμα του ονόματος το οποίο έχει φράξει το δρόμο της ε, χώρας για την προσέγγιση της και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και θα πρέπει να καλύψουμε και το θέμα της ονομασίας της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά, Πρόεδρε. Αυτά για τη συμφωνία που αποσπάσαμε. Ο Πρόεδρος. Ο κύριος Χάουιτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μεγάλη χαρά να μπορέσω να δουλέψω μαζί με τον ε, Έντουαρτ Κούκαν και επίσης και ο της ομάδας ναι. Άλντε ήταν παρόν. Κάναμε ε, πέντε μέρες ουσιαστικά διαμεσολάβησης στο, στα Σκόπια. Μιλήσαμε με τους εμπλεκόμενους όλους προσωπικά και μπορώ να σας πω ότι χρειάστηκε να έρθουμε σε επαφή με όλα τα θέματα της ε, χώρας. Συγγνώμη που δεν ήρθαμε νωρίτερα στην αρχή της διαδικασίας ε, για να παρουσιάσουμε την ε, διαδικασία. Νομίζω ότι μάθαμε πώς να διευκολύνουμε ορισμένες διαδικασίες για την κοινοβουλευτική δημοκρατία και διπλωματία, όπως είπε ο Ed Κούκαν. Κάναμε κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει χωρίς την συμμετοχή κοινοβουλευτικών. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό το γεγονός ότι εμείς μπορέσαμε να λειτουργήσουμε γιατί η κυβερνούσα πλευρά ανήκε στην μεριά του ΕΛΚ και η αντιπολίτευση από την πλευρά των σοσιαλιστών. Μπορέσαμε λοιπόν να τους ε, προσεγγίσουμε μέσω των κομμάτων μας και έτσι να εξομαλύνουμε κάποιες από τις διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ τους. Όλα αυτά δεν ήταν τέλεια, αλλά νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο το να υπάρχει κοινοβουλευτική διπλωματία. Βοήθησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Και νομίζω ότι και ο κύριος Χάνο, αρμόδιος επίτροπος, θα επιθυμούσε την παρουσία κοινοβουλευτικών σε αντίστοιχε περιπτώσεις στο μέλλον και αυτό μπορεί να είναι μια πολύ θετική ε, συμβολή του Κοινοβουλίου. Ο Έντ αναφέρθηκε στις, ε, ε, στο περιεχόμενο της συμφωνίας και νομίζω ότι σωστά δεν ανέφερε τα σημεία που μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω δυσκολίες και διαφωνίες. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια εμπιστευτικότητα για να διατηρήσουμε και την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Τρία γενικά σχόλια. Πρώτον, είναι μια χώρα που έχει μια στη δημοκρατία όπου υπήρξε απόλυτη καταστροφή κάθε μορφής εμπιστοσύνης μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για οποιαδήποτε δημοκρατία. Είναι πολύ αρνητικό για τις προοπτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της χώρας. Και αυτό είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μετά από δύο χρόνια που είχε ήδη καταστραφεί η σχέση των δύο κομμάτων. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο εύθραυστη είναι η δημοκρατία στη χώρα αυτή και σε μερικέ από τι γειτονικέ χώρε που αργά ή γρήγορα θα γίνουν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να είμαστε παρόντες εκεί, να έχουμε την απαραίτητη προσοχή, να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και σκληρή πίεση αν χρειάζεται, αλλά θα πρέπει όλοι να καταλαβαίνουν πόσο δύσκολη, πόσο ευάλωτη είναι η δημοκρατία στη χώρα αυτή και σε μερικές από τις γειτονικέ χώρες. Όταν βγήκαν στη φόρα τα σκάνδαλα, εγώ θεώρησα ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μια επιλεκτική δημοσίευσε από την αντιπολίτευση κάποιων ε, μαγνητοτενιών που δημιούργησε βέβαια κάποια σχόλια. Θεώρησα ότι έπρεπε να συγκρατώ και να μην κάνω σχόλια, αλλά δεν ήθελα να υποστηρίξω μια τέτοια ενέργεια. <clears throat> Πιστεύω ότι το, από ό,τι φαίνεται, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιεχόμενο των ε, ηχογραφήσεων αυτών που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτές μια σειρά από σοβαρά φαινόμενα διαφθοράς και φτάνουν τόσο βαθιά όλα αυτά τα πράγματα ώστε ήταν πιστεύω δικαιολογημένη η χρήση αυτής της τακτικής αλλιώς η κυβερνητική πλευρά δεν θα συμφωνούσε καθόλου για να υπάρξει μια αντιμετώπιση της ε, διαμάχης αυτής. Είναι τόσο σοβαρό λοιπόν το περιεχόμενο των ηχογραφήσεων ώστε απαιτούν το πραγματικά έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Φαίνεται ότι έγιναν 20.000 παρακολουθήσεις παράνομα τηλεφώνων στη χώρα αυτή. Είναι δύσκολο <clears throat> για μας να σκεφτούμε για όλες αυτές τις ε, καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει, αλλά η Κομισιόν έχει μια ομάδα νομικών εμπειρογνωμόνων με ένα επικεφαλής προηγούμενης, προηγούμενο επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης της Κομισιόν και υπάρχει μια έκθεση στο διαδίκτυο που καταγράφει τις κύριες <clears throat> καταγγελίες και για όποιον ενδιαφέρεται για την Ποδογουμού είναι πολύ χρήσιμο να παρακολουθήσει αυτά τα οποία καταγγέλλονται γιατί θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματα τα οποία μπορούν να υπάρχουν σε, σε χώρες όπως η Μακεδονία. Ένα δεύτερο σημείο και εδώ θα προσπαθήσω να επιταχύνω είναι ότι αυτή η συμφωνία δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί αν δεν υπάρχει μεγάλη διεθνής παρουσία και πίεση και στις δύο πλευρές. Φυσικά πρέπει να <clears throat> συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να συζητήσουμε με τους πεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια. Πρέπει πράγματι να ασκήσουμε συνεχή πίεση στα κόμματα για να τηρήσουν μέχρι κεραίας αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι κάτι που συμφωνήσαμε και με τον κύριο Χάν είναι απαραίτητο να υπάρξει πίεση. Θα πάει το Προεδρείο του Κόμματος μας στα Σκόπια την επόμενη εβδομάδα, ίσως και αυτή τη εβδομάδα και θα πρέπει να κάνουμε σαφές ότι πρέπει να τηρηθούν <clears throat> οι δημοκρατικές αρχές. Κανονικά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, αλλά αν γίνεται πρέπει να γίνει προς το συμφέρον όλης της Ευρώπης. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι η απάντηση στο ερώτημα το οποίο έθεσα προηγουμένως στον κύριο Άσελμπρον για τις προοπτικές προσχώρησης. Ο κύριος Χαν έκανε, ανέβ, ανέλαβε ένα ρίσκο όπως και ο κύριος Φίλε όταν είπε ότι θέλει να υπάρξει μια πρόοδος από την Ελλάδα για το θέμα του ονόματος και άνοιγμα συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλοι φραγμοί. Ο κύριος Χαν θεωρεί ότι είναι τόσο ρευστή η κατάσταση στην Αθήνα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για κάποια εξέλιξη η οποία μπορεί να λάβει χώρα το φθινόπωρο και ο Υφυπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν παρόν και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ε, διπλωματική προσπάθεια που έγινε μέχρι χθε και έχει αναφέρει αντίστοιχες προτάσεις για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την συμμετοχή της Μακεδονίας στον ΝΑΤΟ. Εμείς ως Κοινοβούλιο κάθε χρόνο το υποστηρίζουμε αυτό με μεγάλη πλειοψηφία παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας, παρά τα φράγματα που πρέπει, τους πρέπει να ξεπεραστούν. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει μπλοκάρισμα της, ε, εν, της εισδοχής Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, αυτό συμβάλλει και στην ένταση που συνεχίζεται να υπάρχει εκεί. Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα σχετικά ισχυρό μήνυμα από όλους μας για αυτό το θέμα. Κύριε Κούκαν. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, γιατί ο Ρίτσαρτ το είπε. Όντω αξίζει να το πούμε αυτή τη στιγμή ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια επόμενη αντιπροσωπεία υπό τον Πίτερ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή που πηγαίνει εκεί για τις ε, σχέσεις μας με τη Μακεδονία, Τσαμπάσκη και ο Στάνισε από τους σοσιαλιστές πάνε. Θα υπάρχει Προεδρία της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα συζητήσει πώς θα προχωρήσει η συνάντηση αυτή της Επιτροπής για τη Σύνδεση γιατί δεν ήταν δυνατόν να είναι εκτός η αντιπολίτευση. Με αυτή τη νέα κατάσταση τώρα πιστεύω ότι πρέπει υπεύθυνα να συζητήσουν και να χρησιμοποιηθεί αυτή η συνάντηση ως ένα παραπάνω εργαλείο για να υπάρξει έλεγχος επί της εφαρμογής της συμφωνίας. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς? Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την συμβολή της, για τη συμβολή σας κύριε Χάουιτ και κύριε ε, Κούκαν. Πριν από 15 χρόνια θυμάμαι ότι είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο με τα αλβανικά κόμματα, τους επικεφαλείς των αλβανικών κομμάτων που τους είχαμε προσκαλέσει εδώ για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία. Δεν πρέπει αυτός ο οποίος χάνει τις εκλογές να επαναλαμβάνει συνέχεια αυτή τη διαδικασία καταγγελιών και να συνεχίζεται στο ότι είναι και σε αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καταλάβουν όλα τα κόμματα ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένες βασικές συμφωνίες μεταξύ των δύο για να μπορέσουμε να έχουμε μια μονιμότητα και μια βιωσιμότητα στην πολιτική των περιοχών αυτών. Ξέρω λοιπόν ότι ε, πόσο δύσκολα είναι γιατί έχω εμπλακεί και εγώ σε αντίστοιχε διαδικασίε. Όλα αυτά δεν περιορίζουν φυσικά την επιτυχία του εγχείρηματό σα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τελικά θα αυξηθεί η κατανόηση στα κράτη αυτά ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια βιωσιμότητα στην ε, ε, πολιτική των χωρών αυτών. Δεν μπορεί λοιπόν μια παράταξη επειδή είναι στην κυβέρνηση να προσπαθεί να διατηρήσει με κάθε μέσο την εξουσία και μια ιτημένη πλευρά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί την αντιπολίτευση για να ε, ανατρέψει την αντίστοιχη κυβέρνηση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορέσουμε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της... Και σας ε, εύχομαι να μπορέσετε να κοιμηθείτε λιγάκι κύριε Κούκαν και κύριε ε, Χάουτ και καλές διακοπές γιατί το αξίζετε μετά από όλα αυτά που κάνατε και μαζί με τον κύριο Βάγγελ και τον Επίτροπο Χάν που συνέβαλε και αυτή. Έχουμε τώρα το θέμα της Κίνας. Ο κύριος Μπέλντερ θα μας παρουσιάσει τις απόψεις του τώρα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τρίτη φορά που στην Επιτροπή αυτή παρουσιάζω έκθεση για την ε, σημασία που έχουν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Όντως πρόκειται για μεγάλη χώρα και αυτή είναι μεγάλη. Ακριβώς λοιπόν επειδή το θέμα είναι τόσο σημαντικό, οι πληροφορίες πρέπει να είναι και πολιτικές και επιστημονικές. Έχω ένα περιορισμένο κείμενο, έπρεπε να το περιορίσω, γι' αυτό και αναγκάστηκα να κάνω επιλογές και να μην βάλω κάποια πράγματα, τα οποία ελπίζω με τις τροπολογίες να ε, προσθεθούν. Έχουμε 40 χρόνια διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Και όντω υπάρχει μια διπλωματική δυναμική από πλευρά τη Κίνα. Θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εταιρικό ε, εταίρο. Συνεπώ, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της με την Κίνα. Αυτό είναι αναγκαίο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική για να προετοιμαστούν αυτές οι σχέσεις. Τώρα, για να εκτιμήσουμε καλά την κατάσταση, την ε, πολιτική και τις σχέσεις μας με την Κίνα, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η εσωτερική κατάσταση στη χώρα. Στη σημερινή κατάσταση λοιπόν υπάρχει ένας ελκυστικός χαρακτήρας για μια ανοιχτή προσέγγιση προς τον έξω κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και μια καταστολή στο εσωτερικό. Στο ίδιο τμήμα συμπεριλαμβάνω και άλλα πολιτικά σημαντικά ζητήματα. Τις επιπτώσεις, για παράδειγμα, που έχει η εκστρατεία της Κίνας κατά της διαφθοράς, τις οικονομικές ε, επιπτώσεις, την κατάσταση στην κακή όσον αφορά το περιβάλλον στη χώρα. Και αναφέρω βέβαια και το θέμα της τρομοκρατίας που απειλεί όπως την Ευρώπη και την ε, Κίνα το Πεκίνο και όχι μόνο. Και άρα οι συνέπειες είναι μεγάλες κυρίως στην περιοχή του Σινγκιάνγκ. Για την Κίνα τώρα. Να ξέρουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη δύναμη, φυσικά, παγκόσμια. Η σημερινή γεωπολιτική κατάσταση απαιτεί νέα στρατηγική και νέο καθορισμό προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Κίνα. Η εξωτερική κατάσταση τώρα. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την πολιτική της Κίνας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία. Υπάρχουν δραστηριότητες της Κίνας λοιπόν στην Ασία κυρίως και ενισχύει και τις σχέσεις της με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η πολιτική της Κίνας στην νότια συνική θάλασσα επίσης είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Η προσέγγιση του Πεκίνου με την Μόσχα, δεδομένων των σχέσεων που έχει και η Ευρώπη με τον Πούτιν. Έπειτα το θέμα το πυρηνικό. Ξέρουμε ότι η Κίνα μίλησε για τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και οι χώρες μέλη πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο διπλωματικό για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Ένα άλλο τμήμα στην έκθεσή μου είναι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όντω, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Κίνα κάποιε ναι, προσπάθειε. Από την άλλη μεριά, σε ορισμένε περιοχέ επιδεινώνεται η κατάσταση. Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ και την ε, προσπάθεια που γίνεται από πλευρά τη ε, Κίνης για κινεζοποίηση θρησκεών του χριστιανισμού για παράδειγμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσουν σίγουρα και ελπίζω με τροπολογίες να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτό το θέμα. Τέλος, για τις σχέσεις της Κίνας με την Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι η Ταϊβάν μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Βοηθάει στη σταθερότητα στην περιοχή και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει η Ταϊβάν προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, συνάδελφοι, με τους κοιόδης συζητητές είχα καλή συνεργασία και του ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα περιμένω τι δικέ σα παρατηρήσει τα σχόλιά σα, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή και να στείλουμε ένα καλό μήνυμα για τη σχέση μας με την Κίνα, η οποία Κίνα έχει τεράστιο δυναμικό το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να συνεργαστούμε καλά, γνωρίζοντας όμως και περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να παρουσιάσω την θέση του συναδέρφου Λόπες που είναι σκιώδης. Εισηγητής αλλά δεν είναι εδώ τώρα. Ετοίμασε στα αγγλικά κάτι και θα σας το διαβάσω λοιπόν και εγώ στα αγγλικά. Ε, Σκέφτεσαι εισηγητής ευχαριστεί τον κύριο Μπέλτερ Θεωρεί ότι η έκθεσή του είναι καλή βάση για να δουλέψουμε πάνω σε αυτή. Θα εμπλουτιστεί με σε κάποια σημεία του κειμένου. Κάπου θέλει επαναδιατύπωση κάποιων ιδεών για τα εξή. Πρώτον, για το αποτέλεσμα της τελευταίας διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας που αναφέρεται και στη στρατηγική συνεργασία για το 2020. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία και να ενισχυθεί η εταιρική σχέση μεταξύ τους. Δεύτερον, οι συνεχιζόμενες συμφωνίες για επενδύσεις έχουν τεράστια ε, σημασία. Δεν είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής, αλλά οι πολιτικές επιπτώσεις μιας τέτοιας συμφωνίας <laughs> πηγαίνουν πέρα από την οικονομική διάσταση. Τρίτον, η κατάσταση στην νότια συνική θάλασσα και οι προκλήσεις που γίνονται από τις διάφορες πλευρές εντείνουν τις δυσκολίες. Άρα χρειάζεται ένας μηχανισμός διαχείρισης αυτών των εντάσεων. Ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες και όχι μόνο τοπικές. Γι' αυτό πρέπει να διευθετηθεί το θέμα της ε, κυκλοφορίας στην περιοχή και να ενισχύσουμε αυτή την παράγραφο που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα στην Νότια Συνική Θάλασσα. Έπειτα, ε, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε συντονισμό με τις Ηνωμένε Πολιτείες, πολύ σημαντικό, αλλά επιπλέον θα ήθελε ο Σκέφτης συγκεκριτής να καταλάβει καλύτερα τι εννοεί στην παράγραφο 10 ο η συγητής, ο οποίος μιλάει για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ε, την Ασία σε διατλαντικό πλαίσιο. Επίσης, ίσως δεν κατάλαβε καλά τον ε, εισηγητή, αλλά πιστεύει ότι η στρατηγική μας για την Κίνα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια ε, της συνεργασίας και ανταγωνισμού. Επίσης, θέλει να λάβουμε υπόψη μας το θέμα της ασφάλειας, που από αντιλαμβάνεται δεν εξετάζεται παρκώς εδώ. Επειδή υπάρχει το θέμα της επικοινωνίας των ε, κινέζικων αρχών και επίσης πρόσφατα η Κίνα αποφάσισε για την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο. Είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε δελεχέστερα. Επίσης, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ίσως στην παράγραφο 17 να μπορούμε να συμπληρώσουμε κάτι. Σίγουρα πρέπει να ελέγξουμε τι θα γίνει με τον κύριο Λεμπρινίδη που θα πάει στην Κίνα και να παρακολουθήσουμε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε δύο θέματα που θα εξεταστούν στην διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι και στη διάσκεψη για την Ατζέντα 2015 στην συνέλευση του ΟΙΕ. Πρόκειται για δύο καλές ευκαιρίες ώστε εκείνο να αποδείξει τον κόσμο ότι μιλάει σοβαρά όταν λέει ότι θέλει να είναι ένας διεθνής εταίρος. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω και εγώ δύο λόγια για το θέμα του Θιβέτ. Γιατί όπως διαβάσαμε πριν από λίγο καιρό, ο Τενζίκ Τελέκυπος πέθανε σε μια κινέζικη φυλακή το 2002 είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ζήτησε να απελευθερωθεί. Κάθε φορά που υπήρχαν συνομιλίες με την Κίνα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι και αυτό και αυτοί οι υπερπολισμοί στο Θιβέτ έχουν οδηγήσει σε 140 τέτοιες περιπτώσεις από το 2009. Η έκθεση λοιπόν αυτή για την Κίνα αποτελεί μια ευκαιρία για να επαναλάβουμε το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Θιβέτ. Δεν πρέπει να διαφορούμε για το Θιβέτ, αντίθετα πρέπει να τολμήσουμε να το θέτουμε στις σχέσεις μας με την Κίνα. Κυρίως μάλιστα που τώρα η Κίνα αρνείται κάθε διάλογο με το Δαλάη Λάμα. Πρέπει να υπάρχει τέτοιος διάλογος. Οι τελευταίες συνομιλίες ήταν το 2010 και δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόοδος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να στοιχηματίσει για την επανάληψη των συνομιλιών. Γιατί μόνο τότε οι Θηβετιανοί θα είναι ελεύθεροι να σκίσουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Λάινεν. Ο κύριος Λάινεν. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μου πλευρά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέλντερ για το σχέδιο της νέας αυτής έκθεσης για την Κίνα. Κυρίως γιατί έχει ήδη για τις επαφή με τους κοιόδης συζητητές και κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Η αντιπροσωπεία για την Κίνα θα ταξιδέψει την Κυριακή, θα πάει την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο και στο Σινκιάν και αυτά τα οποία πρέπει να συζητηθούν και οι δικέ μας θέσεις που πρέπει να παρουσιάσουμε έναντι των εταίρων μας στην Κίνα. Ο κύριος Μπέλντερ αναφέρθηκε και στην έκθεση Μογκερίνη η οποία θα ακολουθήσει το φθινόπωρο και θα περιλαμβάνει μια νέα στρατηγική για την Κίνα. Πιστεύω ότι και η δική μας έκθεση θα πρέπει να δώσει κατευθύνσεις στην Κομισιόν για να γίνει σαφές τι θέλουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Η στρατηγική σκέψη, σχέση μάλλον, θα πρέπει να αναφερθεί ως πρώτο κεφάλαιο στην έκθεση κατά τη δική μου άποψη. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα με τις εσωτερικές συνθήκες στην Κίνα. Έχουν οριμάσει οι σχέσεις μας. Η Κίνα είναι μια μεγάλη δύναμη ένας ε, σημαντικός παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα έχουν πολλά κοινά εγχειρήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Επομένως αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και περισσότερο και στην έκθεση αυτή. Η παγκόσμια διακυβέρνηση, η, η... Ε, η επίτευξη της ειρήνης και διατήρησή της, οι σχέσεις με το Ιράν, με τη Συρία, με την Ουκρανία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να συμβάλλει και η Κίνα στα εγχειρήματα αυτά. Ε, αναφέρεται επίσης η πολιτική για τα κλιματικά θέματα. Ξέρω ότι έμαθα ότι η Κίνα θα δημιουργήσει ένα δικό της ταμείο για την κλιματική αλλαγή, ένα πράσινο ταμείο. Και αναρωτιέμαι τώρα γιατί η Κίνα θέλει να δημιουργήσει ανεξάρτητα εργαλεία και φορείς και δεν θέλει να συμβάλλει στους πολυμερείς φορείς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που υπάρχουν ήδη. Επίσης, το θέμα του, των εμπορικών ζητημάτων και οικονομικών ζητημάτων, εγώ πιστεύω πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά στις επενδυτικές συμφωνίες, το καθεστώς της οικονομίας αγορά αγοράς στην Κίνα, το θέμα της συμμετοχής της Κίνας στους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτή την έκθεση. Για τα θέματα της εσωτερικής πολιτικής της Κίνας, προφανώς μας ανησυχεί το επίπεδο καταστολής, η περιπτώση καταστολής που έχουμε δει στην Κίνα. Δεν μπορεί να είναι μια εξέλιξη την οποία μπορούμε να επικροτήσουμε, ούτε ο νόμος για τις ΜΚΟ, ούτε ο νόμος για την ασφάλεια που έχει μια πάρα πολύ ευρεία έννοια της ασφάλειας που διεισδύει σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της ανθρώπινης ζωής, η έλλειψη κράτους δικαίου και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολίτες στην Κίνα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, περιληφθεί στην έκθεση και δεν θα πρέπει να έχουμε να διστάσουμε να τα αναφέρουμε αυτά. Επίσης η σύγκρουση στο νότιο συνικό πέλαγος και εκεί θα πρέπει να συμβάλλουμε σε την επίτευξη μιας πολιτικής λύσης και όχι σε μια αντιπαράθεση σε στρατιωτικό επίπεδο. Πιστεύω ότι η Κίνα θα πρέπει να παίξει ένα, ένα οικοδομητικό ρόλο επίσης και σε σχέση με την προβληματική της Βόρειας Κορέας. Και επίσης ο εισηγητής έχει αναφερθεί και στην ανακατεύθυνση των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Ρωσίας το αν υπάρχει μια τέτοια συνεργασία η οποία αν αυτή η συνεργασία καλύτερα στρέφεται εναντίον μας ή είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να μπορέσει να συμμετάσχει στην κοινή αυτή συνεργασία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης. Υπάρχει πίεση κατά των ε, θρησκευτικών ομολογιών, όχι μονάχα της χριστιανικής θρησκείας αλλά και άλλων ε, δογμάτων. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Υπάρχει λογοκρισία στο διαδίκτυο οι ξένες ε, αλλά και οι εγχώριες ΜΚΟ έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Το Θήβετ ισχύει εκεί όπως και στο παρελθόν καταστολή οι σχέσεις με την Ταϊβάν. Ίσως πρέπει να επενέσουμε το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί αυτές οι σχέσεις. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει να εκφράσουμε την ε, λύπη μας για το γεγονός ότι η Κίνα έχει ενισχύσει τον νόμο περί μη αποσχήσεως και προβλέπει να χρησιμοποιήσει ακόμα και στρατιωτικά μέσα για να τα αντιμετωπίσει μια τέτοια δεχόμενη απόσχηση. Δεν βλέπω να αναφέρεται κάτι για το Χονγκ Κόνγκ εδώ. Το θέμα της ε, εκλογής του ανώτατου εκτελεστικού άρχοντα που θα είναι πηγή συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί, θα πρέπει να κάνουμε μια έκκληση και προς δύο πλευρές να βρουν συμβαστικές λύσεις και όχι να οξύνουν ακόμα περισσότερο την ε, διαμάχη αυτή και να οδηγηθούν σε αντιπαραθέσεις βίες. Έχω να, καταθέσει, έχω να καταθέσω κάποιες τροπολογίες που πιστεύω ότι θα παρουσιάσουν με αντικειμενικό ε, τρόπο την κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση και ίσως είναι μόνη τέτοια έκθεση για την Κίνα την τρέχουσα νομοθετική περίοδο θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε το δρόμο προς το 20, 2020 σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα. Ευχαριστώ. Φαντάλεν. Be reminded 10 minutes the high rep will be here. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ η, η πάτη εκπρόσωπος. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουμε η έκθεση του κυρίου συναδέλφου είναι πάρα πολύ αξιόλογη Απλώς θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο τα θέματα τα εμπορικά. Ήδη περιλαμβάνονται εδώ, αλλά θα πρέπει, αν και δεν πρόκειται περί δημοκρατίας, με τίποτα δεν τους λέω ότι είναι δημοκρατία, ούτε κανένα διόμενη δημοκρατία, αλλά θα πρέπει ακριβώς, επειδή έχουμε αυτήν την τεταμένη σχέση με τη Ρωσία, θα πρέπει να κοιτούμε προς την Κίνα, ακριβώς όπως έχει κάνει και η Αμερική. Άρα να επικεντρωθούμε περισσότερο στην, ε, στην εμπορική δραστηριότητα. Είναι βέβαια μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και άρα θα πρέπει ε, να δούμε πώς θα ε, εμπλακεί σε όλα τα φόρα, σε όλες τις διεθνείς ρυθμίσεις της εμπορικές εκείνα Τώρα άλλα δύο ζητήματα που θέλω να δείξω. Πρώτα πρώτα το Χογκόνγκ. Το Χογκόνγκ είναι αυτόνομη περιφέρεια όπως γνωρίζουμε. Όμως ο λαός εκεί δεν μπορεί να εκλέξει τον κυβερνήτη του, chief executive. Δεν ξέρω από την ε, Κίνα. ...αλλά θα πρέπει εμείς αυτό να προωθήσουμε, να δικαιούται ο λαό να εκλέξει τον chief executive, τον κυβερνήτη. Ε, τώρα, θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι εμείς θέλουμε να ισχύσει το status quo όσον αφορά στις σχέσεις με την Ταϊβάν. Η Κίνα τους θεωρεί σαν ε, ε, μια επαρχία σε κατάσταση ανυπακοής και παρανομίας, αλλά εμεί θα πρέπει για όλα τα εμπορικά θέματα να προωθήσουμε ότι θα πρέπει να ισχύσει το στάθος του να υπάρξει επίσης ε, μια αναθεώρηση του κειμένου, να κάνουμε συνεργασία περισσότερο για την υψηλή τεχνολογία, γιατί οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ καλή στο να ε, έχουν τη μεταδρομή, το μετασχηματισμό τέλο πάντων από το υλικό, το χίδιν υλικό σε υψηλή τεχνολογία. Ο επόμενο κύριε Μίκη. Άκουσα πρόεδρε ότι με, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και χέρι-χέρι με τους Αμερικανούς θα πιέσουμε την Κίνα. Αλλά το άκουσα αυτό θα γίνει και με την Ρωσία. Αλλά το μόνο αποτέλεσμα είναι ότι έτσι την συμμαχία, την Ρώσο-Κινέζικη την κάνετε πιο ισχυρή και συγχαρητήρια. Μα τι θέλετε να, ε, να αναμειχθούμε στις διεκδικήσεις για τις κουρίλες και τις άλλες αυτές διεκδικήσεις. Μιλάν μόνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Κατά τη γνώμη μου αυτή η έκθεση αναφέρει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι σχέσεις με την Κίνα που είναι πάρα πολύ σημαντική, αναδυόμενη δύναμη, πάρα πολύ βασικό θέμα της τελευταίας 20 αιτίας. Και από την άλλη μεριά νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι κάπως διστακτική, κάπως αμυντική, οίκιστα φιλόδοξη και θετική. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τη σχέση μας με την Κίνα με πιο πολύ θετικό πνεύμα. Οπότε και εγώ θα επεξέτεινα κάπως παραπάνω τις πρώτες τρεις παραγράφους. Στρατηγική, πολιτική, συνεργασία κλπ. Όλα αυτά τα σχετικά ε, χρειάζονται κάπως ε, ε, επέκταση. Να γράψουμε περισσότερα. Μα τι λέμε εδώ πέρα, λέμε μόνο στην τρίτη μόνο για το ISDS, μα οι σχέση μας με την Κίνα είναι πολύ παραπάνω από αυτή τη διαδικασία Και πριν από δύο-τρει εβδομάδε είχαμε αυτή τη συνάντηση κορυφή με τη χώρα εκείνη, όπου νομίζω ότι προέκυψαν πάρα πολλά. Είναι τόσο σημαντικό παίκτη η Κίνα στον ε, πολυπολικό αυτόν κόσμο και επομένω θα πρέπει εμεί να μην παρεπιοριστούμε σε αυτά. Θα πρέπει να αναδείξουμε όλε τι θετικέ πλευρέ τη σχέση. Γιατί επομένω αυτό λείπει από εδώ. γιατί κατάφεραν να καταπονήσουν την ε, Κίνα, υπάρχει μια ολόκληρη αντιομενιστική τάξη εκεί, ε, θα πρέπει να πούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, τα βήματα πρώτα που εσημείωσαν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι φαινόμενο του 20ου αιώνα, από τη δεκαετία του 90 και μετά τουλάχιστον, άρα πέστε τα πιο θετικά παρακαλώ. Και επίσης για τη στρατηγική μας. Είμαστε μία 28 χωρών, η Κίνα είναι ένας γίγαντας σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο ε, και θα πρέπει εμείς πέραν της σχέσης με τη ΣΥΠΑ να φροντίσουμε και τη σχέση μας με την Κίνα. Ας τα λέμε, ας συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς αλλά θα πρέπει να μην εξαρτάται η σχέση μας με την Κίνα από τους Αμερικανούς. Α, αυτές είναι οι σκέψεις μου. Αλλά επιμένω, πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Και επομένως θα πρέπει και εμείς με την έκθεσή μας να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων της σημασίας του θέματος. Μποστινάρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ αρχίζω λέγοντας το πώς το είμαι στο ίδιο μήκο κύματο με τον συνάδελφο του ΕΛΚ, τον κύριο Μιλιάν Μον. Γιατί οι, οι εκθέσει μα θα πρέπει να εξυπηρετούν τι γεωστρατηγικέ σχέσει με την Κίνα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, θα πρέπει να είναι δίκαιε οι γνώμε εκεί και κυρίω θα πρέπει να είναι ρεαλιστικέ οι εκθέσει. Και έτσι η Ευρώπη να μπορεί να χαράξει καλύτερα τη στρατηγική με την Κίνα και θα πρέπει επίσης να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στατική σχέση. Άρα κατά την ταπεινή μου γνώμη, τι λείπει από εδώ πρώτον για το περιβάλλον. Καλά, λέμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά όπως είπε και ο Μπέλντερ, ο Λόρδος Τέλιν, ο Λόρδος Τέλιν, ο οποίος ε, εκτιμάται τόσο πολύ, συνέντευξε αυτή την έκθεση στο London School of και είπε για την ε, πρόοδο της Κίνας στο μέτωπο του περιβάλλοντος. Ότι είπε πως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η πρόοδος και ότι ήταν συνεπής η Κίνα σε σχέση με τις υποσχέσεις. Μα αυτό μπορεί να το αγνοήσουμε. Ε, έχουμε αυτή την κοινή δήλωση επίση. Πριν από δύο εβδομάδες την συνεπογράψαμε με την Κίνα. Για πρώτη φορά η Ευρώπη και η Κίνα ε, δεσμεύτηκαν από κοινού εν ώψη της διάσκεψης των Παρισίων. Για πρώτη φορά συνυπογράψαμε κάτι για το περιβάλλον. Μα είναι δυνατόν να μην το αναφέρουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη στρατηγική μας. Και επίσης Κίνα και Ευρώπη είπαν ότι θέλουν να εργαστούν εν ώψη της διάσκεψης της Αντίσα για την ανάπτυξη. Και αυτό είναι σημαντικό για μας, για τους στόχους μας δεν πρέπει να το αναφέρουμε. Ε, βέβαια και πρέπει. Επίσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποιος είναι ο ρόλος της Κίνας στο ταμείο αυτό. Ίσως ξέρουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα ε, ένα γραφείο, μια αποστολή τέλος πάντων του Δουνουτού και τώρα θέλουν να ζυγίσουν το μήπως το Ιουάν, το νόμισμα το, το Κινέζικο θα πρέπει να μπει στο καλάθι του, του του. Μα δεν είναι σημαντικό αυτό. Φυσικά και είναι και πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση. Πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά την διμερή συμφωνία, είναι σημαντικό να πούμε το τι προσδοκούμε από την επενδυτική συμφωνία, να πούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, αλλά επίσης να πούμε το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις αφού εγκριθεί το ψήφισμα για το TTIP. Το οποίο είναι σίγουρο ότι θα περιέχεται στη συμφωνία, γιατί ίσως δεν το ξέρετε, αλλά ίσως για, στο TTIP να συμμετάσχει κάποια στιγμή η Κίνα και κάποια στιγμή επίσης οι ΙΠΑ να προσχωρήσουν στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης. Ε, δεν θα πρέπει όλα αυτά να αναφερθούν. Ε, βέβαια. Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τα βασικά στοιχεία της ε, συνάντησης κορυφής Κίνας ΕΕ. Και, ε, κάτι είπε ο κύριος Μίκη, εκτός Μπετίνη. Πηγαίνει ο χρόνος, οπότε και θα, θα, ήθελα να πω και κάποια ε, γενικόλογα σημεία, αλλά γιατί το είπαν και οι συνάδελφοι, αλλά εγώ δεν με κάλυψαν συνάδελφοι, οπότε θέλω να αναφέρω μόνο τα εξή. Πρώτον, όσον αφορά το Θιβέτ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαλαρή η διατύπωση, πάρα πολύ ήπια, θα πρέπει να την κάνουμε πιο δυναμική. Ακριβώς όπως είπαμε και για το Βιετνάμ. Επίσης, πώς θα μπορέσουμε να εξοφίσουμε την Κίνα να κάνει βήματα πρόοδου να ακολουθήσει το μονοπάτι της οικονομίας της αγοράς που δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει τώρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να το θίξουν. Σε μισό λεπτό θα είναι εδώ. Ε, Danke, Herr Äh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο, Πολλά υπόθηκαν ήδη. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση δεν πηγαίνει αρκετά μακριά. Γιατί μιλάει πολύ για τις δυσκολίες, για τις κοινέ προκλήσεις. Και έχοντας ακούσει και τον συνάδελφο Μποστινάρο και τον συνάδελφο Λάινεν, θα έλεγα και εγώ ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο το θέμα της ε, στρατηγικής συνεργασίας για ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να συνεργαστούμε με την Κίνα. Πρόκειται για τρίτε εκατομμύρια ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τι κατανάλωση σημαίνει αυτό. Τρόφιμα, ανθρώπινα δικαιώματα, ό,τι γίνεται στην Κίνα μας αφορά. Αυτό θέλω να πω το αν η Κίνα πετύχει ή αποτύχει, αυτό έχει αντίκτυπο σε εμά, στη δικιά μας τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με την Κίνα με άλλους. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε κάπως την προσέγγισή μας. Πιστεύω ότι η Κίνα είναι στρατηγικός εταίρος. Πρόεδρος. Ωραία. Ο κύριος Λάινεν χαίρομαι που είπε ότι θα υποβάλει τροπολογίες ήπιες και αντικειμενικές. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Πάντως το μόνο που θέλω τώρα να ζητήσω από τον εισηγητή είναι μήπως θα μπορούσε να προσθέσει ένα πράγμα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, γιατί είναι μια οικονομία της αγοράς η Κίνα, αλλά όλα όσα έχουν να κάνουν με τις λεπτομέρειες της αγοράς αυτής περνούν από το κράτος. Υπάρχει αυτή η συνολική στρατηγική της Κίνας, υπάρχει η πολιτική άμυνας, όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια μιας συνολικής στρατηγικής. Αλλά τι γίνεται με μια εντελώ ελεύθερη οικονομία. Δεν είναι η περίπτωση της Κίνας βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι στο σύστημα υπάρχουν ε, εντάσεις. Μήπως λοιπόν θα μπορούσατε πριν ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή να μας το διευκρινίσετε κύριε Μπέλντερ και παρακαλώ να είσαστε σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την ιδέα. Σας είπα ότι άφησα πολλά πράγματα έξω από την έκθεση αυτή. Τα οικονομικά ζητήματα για παράδειγμα, αλλά και άλλα. Εντάξει, οι τροπολογίες και ίντα και άλλοι μπορούν να υποβάλουν. Υπάρχει ένα θέμα που είναι αξιοσημείο εδώ. Έφυγε ο κύριος Μποστινάρου βέβαια. Το London School of Economics είχε διαφορετική άποψη. Εκπλήσει. Κοιτάξτε, νομίζω στην έκθεση για την Κίνα πρέπει να δούμε τι λέει η ίδια η Κίνα και να είμαστε επικριτικοί βέβαια. Αλλά πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και ισορροπημένοι. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ποια είναι η θέση των Κινέζων και ποια είναι η θέση δικιά μας. Είναι, πώς να το πω, δουλειά που συνεχίζεται. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις τροπολογίες σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλντερ. Λοιπόν, σας εύχομαι καλές διακοπές. 31 Αυγούστου θα τα ξαναπούμε και ελπίζω να είσαστε σε φόρμα. Καλές διακοπές σε όλους.